Yes, ladies and gentlemen, and first of all, I'd like to... Κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα θερμά να σας καλωσορίσω εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια της ε, διακοινοβουλευτικής συνάντησή μας για το μέλλον της ε, περιφερειακής πολιτικής μετά από το 2013. Ε, καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη ε, εξ ονόματος του Προέδρου της Επιτροπής μας, ο οποίος επιγόντως προσεκλήθη από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ε, και δεν θα μπορέσει να είναι εδώ εξ αρχής, θα έρθει αργότερα. Ο κύριος Γαλεώτη θα έρθει κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Και θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Τσεχικής Δημοκρατίας ε, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, τον κύριο Χορτσίσκα, τον κύριο Ιβο Μπάρεκ που είναι πρόεδρος ε, της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ε, Τσεχικής Γερουσίας, την κυρία Μαρή Βέιμελ Κόρνιας που είναι μέλος της ε, Επιτροπής ε, Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Έχουμε εκπρόσωπο δηλαδή και της μελλοντική Προεδρίας, της Σουηδικής εδώ και βεβαίως ε, τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, τον κύριο Ντεχάνε. Καλώς ορίσατε λοιπόν όλοι και Όλοι θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Θα ήθελα καταρχήν να σας δώσω κάποιες πρακτικές φύσεις ε, πληροφορίες σε σχέση με τη συζήτησή μας. Πρώτον, η αναλογία ανάμεσα στους ομιλητές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι δύο προς ένα, δηλαδή δύο μέλη ε, Εθνικών Κοινοβουλίων και ένα μέλος της Επιτροπής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε και θα θέλαμε να ζητήσουμε εντόνως οι εισηγήσει να μην υπερβαίνουν τα τρία λεπτά πάνω κάτω. Υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις στα εθνικά κοινοβούλια. Η παράδοση εδώ είναι τρία λεπτά θεωρείται πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το τι ήθιστε. Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ να συμπληρώσει αυτό το δελτίο που έχετε, μέσω του οποίου μπορείτε να ζητήσετε το λόγο. Οπότε, παρακαλώ να συμπληρώσετε αυτό το δελτίο και εμείς θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε έτσι τη συζήτηση. Δύο εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, ένας του Ευρω... της Ευρωβουλής. Θα βρείτε το δελτίο αυτό στους φακέλους σας, μέσα σε αυτό το φάκελο που έχετε μπροστά σας. Υπάρχει αυτό το δελτίο. Η συζήτησή μας θα συνεχιστεί μέχρι τις 5.30. Πάνω κάτω. Αν χρειαστεί, μπορεί να πάμε και λίγο παραπάνω. Να σας δώσω και μια πληροφορία σε σχέση με αυτού του είδους ε, τις εργασίες που έχουμε ήδη κάνει στην Επιτροπή μας. Και τώρα θα μιλήσω στη γλώσσα μου, στα πολωνικά δηλαδή, γι' αυτό βάλτε όλα τα ακουστικά σας. Θα ήθελα να πω πόσο σημαντική είναι αυτή η χρονική στιγμή για όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και κυρίως για την πολιτική συνοχής. Η συζήτηση που έχουμε σήμερα γίνεται σε μια φάση όπου ταυτόχρονα εκπονείται και η ενδιάμεση έκθεση, αναθεώρηση και επίσης διαγράφεται το πλαίσιο ε, για την ε, πολιτική συνοχή μετά το 2013. Κανεί δεν ήξερε όταν είχε προγραμματιστεί αυτή η συζήτηση ποιο θα είναι το πλαίσιο. Υπάρχουν ε, οικονομικές δυσκολίες αυτή τη στιγμή που σημαίνουν ότι πολιτική συνοχή και η σχετική συζήτηση θα διαφέρει από αυτό που ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν θα συζητήσουμε πλέον μόνο για την καλύτερη εφαρμογή αυτής της πολιτικής συνοχή, αλλά και για το τι είδο πολιτική συνοχή χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στα επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου γίνεται πολύ σοβαρή συζήτηση όσον αφορά την ίδια την ε, ουσία αυτής της πολιτικής. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας συνέταξε ένα ολόκληρο πακέτο, μια δέσμη κανονισμών για το 2007 μέχρι 2013. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για την μεταρρύθμιση αυτού του πακέτου και πρόκειται για μια εξαιρετική κατάσταση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περίοδου να βλέπουμε τροποποιήσεις στους κανονισμούς. Έχουμε λάβει προτάσεις από το Συμβούλιο επί τη βάση προτάσεων της Επιτροπής και αυτή τη στιγμή εμείς διατυπώνουμε τις απαντήσεις μας προς τις προτάσεις αυτές. Το θέμα αφορά και τα 27 κράτη-μέλη και η συζήτησή μας γίνεται με βάση τις σημερινές αλλαγές στην πολιτική συνοχή. Δηλαδή, οι αλλαγές που γίνονται τώρα στην πολιτική συνοχή θα έχουν συνέπειες και για την περίοδο μετά το 2013. Δηλαδή, οτιδήποτε αλλάξουμε τώρα θα προαναγγέλει το τι θα γίνει μετά το 2013. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας κυρίες και κύριοι σε κάποια θέματα κλειδιά που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Καταρχήν το θέμα του ρόλου αυτής της πολιτικής και η σχέση της με άλλες κοινωτικές πολιτικές. Ποια είναι η προσθήκη συμβολή αυτής της πολιτικής και ποια θα είναι η θέση της στο προπολογισμό για το μέλλον. Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα, αλλά φυσικά πολλά θα εξαρτηθούν από το πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής και τους στόχους της για τα επόμενα χρόνια και έτσι έρχομαι και στο θέμα, στο ερώτημα του τι επιθυμούμε να καλύψουμε με τις δαπάνες της πολιτικής συνοχής. Θέλουμε να δαπανίσουμε χρήματα μόνο για αυτά που χρειάζονται οι φτωχότερες χώρες και περιφέρειες, δηλαδή για τις υποδομές, ή θα πρέπει τα χρήματα να δαπανηθούν και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ε, δηλαδή για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, όπως αποκαλούνται, καινοτομία, ενίσχυση των κέντρων αριστείας. Με άλλα λόγια, αυτή η πολιτική θα είναι μόνο μια πολιτική που θα αφορά τις θεμελιώδεις υποδομές της Ευρώπης ή θα πρέπει να μετατραπεί σε μια ευρύτερη πολιτική που θα καλύπτει ένα σωρό Και έτσι έρχομαι και στο επόμενο ερώτημα. Θα πρέπει να είναι μια πολιτική για τις στοχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα πρέπει να είναι πολιτική για όλες τις περιφέρειες της Ένωσης δεδομένου ότι πιθανότατα θα υπάρξει διαφοροποίηση σε σχέση με τους στόχους. Κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη ότι ορισμένα κράτη-μέλη, όπως ίσως τα γνωρίζετε, ήδη είναι της άποψης ότι δεν χρειάζεται καν να υπάρχει ο στόχος 2 στο μέλλον. Δηλαδή θα μας μείνει μόνο ο στόχος 1. Ε, Επίση ακούσαμε την πρόταση για επανεθνικοποίηση τμήματος αυτής της πολιτικής. Να επιστραφεί δηλαδή η αρμοδιότητα αυτή στα, στις κυβερνήσεις και να δοθούν και κάποια από τα χρήματα που έχουν ε, ε, προβλεφθεί για αυτές τις πολιτικές της ε, κυβερνήσεις. Δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσει να είναι μια πραγματικά κοινοτική πολιτική ή θα πρέπει να είναι και εθνική ε, πολιτική. Δηλαδή όχι μόνο πόσα αλλά και για ποιο σκοπό και από ποιον. Μια απάντηση προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, έχει προέλθει από μια, ε, ένα είδος συνεργασίας μέσα στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας, δηλαδή περιφερειακή και κοινωνική ε, συνοχή. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει αυτή τη στιγμή διαβούλευση με τη μορφή του πράσινου βιβλίου που έχει εκπονήσει για το θέμα. Η περιφερειακή συνοχή δεν είναι μόνο μια νέα διάσταση, αλλά αποτελεί και μια νέα προσέγγιση στην ε, πολιτική συνοχή. Μια νέα προσέγγιση που βασίζεται στην ιδέα της εξισορρόπησης των ευκαιριών που δίνονται στις διάφορες ε, περιφέρειες και είμαι βέβαιος πως κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, θα το ακούσουμε αυτό, καθιστά δυνατή την υποστήριξη για διάφορα είδη περιφερειών, μεγάλες περιφέρειες, μικρές πόλεις και ακόμα και ολόκληρες ομάδες χωρών να αναφέρω μόνο την στρατηγική της Βαλτικής ως παράδειγμα. Κυρίες και κύριοι, για τη Εθνικά Κοινοβούλια η εδαφική συνοχή ανέκαθεν ήταν κάτι που θεωρείται ως κάτι παραπάνω από ένα νέο σύνθημα, αλλά ως μια πρόταση για αλλαγή της ίδιας της φύσης της πολιτικής συνοχής. Εμείς έχουμε εδώ εκπονήσει διάφορες εκθέσεις ε, στον τομέα αυτό. Η μία είναι του κυρίου Γκέλεκ για το τέταρτο, την τέταρτη έκθεση για την πολιτική συνοχή, μια ανέκθεση για την ε, περιφερειακή ατζέντα ε, από την, που την έχει συντάξει η κυρία Κάλεμπαχ. Η Επιτροπή μας έχει συντάξει έκθεση για το θέμα της εταιρικής σχέσης και την ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με εισηγητή τον κύριο Μποπουή και επίσης έχουμε την, την ε, δαφική συνοχή, την ε, έκθεση την οποία έχει συντάξει ο κ. Βανίστελ. Θα ακούσετε πολλούς από όσους ανέφερα απόψε η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Επιτροπή μας και μέσα στις πολιτικές ομάδες που αντιπροσωπεύονται στην Επιτροπή μας. Είναι πολύ σημαντική χρονική στιγμή, συγκυρία, είναι μια σημαντική καμπή. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ πολύ σημαντικές και για να σας μιλήσω για πολιτικούς όρους έχουμε ακόμα δύο μήνες μονάχα στη θητεία μας. Ε, γνωρίζουμε ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση και πρέπει τώρα τώρα να ε, ε, γίνει αυτό. Δεν έχουμε άλλο καιρό να περιμένουμε και γι' αυτό και προσβλέπουμε στην ενεργή σας συμμετοχή. Θα ήθελα λοιπόν κυρίες και κύριοι αυτή τη στιγμή να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Υπουργού τη Εχικής Δημοκρατία για την υπεύθυνο για την ανάπτυξη, του κύριο Χόρετζακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση από την Επιτροπή Ρέτζη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του Υπουργού που για πολύ σοβαρούς λόγους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα εδώ. πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η συζήτηση για, το, για τη μελλοντική διαμόρφωση της πολιτικής συνοχής θα επηρεαστεί από τις οικονομικές εξελίξεις στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι το πρόγραμμα της Τσεχικής Προεδρίας και οι προτεραιότητες ε, της Τσεχικής Προεδρίας για τούτο το εξάμεινο έχουν ε, επηρεαστεί από εξωτερικά γεγονότα και συνθήκες. Όπως ε, θα ακούσατε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται πάνω σε ένα πακέτο νομοθεσίας ε, που σκοπό έχει να τροποποιήσει τους εφαρμοστικούς κανονισμούς κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο. Ωστόσο, δεν θέλουμε να ξεφύγουμε τελείω από έναν από του βασικού στόχου τη Τσεχική Προεδρία, που είναι μια δημόσια συζήτηση για την ε, πολιτική συνοχή. Και άλλωστε, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Η Τσεχική ε, Δημοκρατία θέλει να συνεχιστεί η συζήτηση για την παρούσα στρατηγική και τι ε, προτεραιότητε και για το εάν αντικατοπτρίζουν τους πραγματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η πολιτική για να ανταποκριθεί στις παρούσες προκλήσεις. Υπό τις συνθήκες αυτές η Τσεχική Προεδρία σκοπεύει να συνεχίσει την συζήτηση για την απλοποίηση των εφαρμοστικών κανόνων. Άλλη προτεραιότητα της Τσεχικής Προεδρίας αυτή τη στιγμή είναι η συνέχιση της δημόσιας συζήτησης για την εδαφική συνοχή. Θα θέλαμε να διαβρύνουμε τη συζήτηση αυτή, να διαβρύνουμε το πεδίο της συζήτησης αυτής για να καλύψουμε εκδηλώσεις όπως η παρούσα και άλλες εκδηλώσεις ε, που οργανώνει η Τσεχική Προεδρία που στόχο έχουν να μας ε, δώσουν ε, το υλικό που χρειαζόμαστε μέσω αντιδράσεων μέχρι ε, κριτικών της πολιτικής αυτής. Ε, περιμένω να ακούσω τα θέματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής. Κάποια από αυτά ε, τα έχει ήδη αναφέρει ο πρόεδρος πολύ σωστά. Εγώ προσωπικά, εκ μέρους της Τσεχικής Δημοκρατίας, θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις απαντήσεις αυτές και η Τσεχία θέλει να λάβει υπόψη της τα όσα θα υποθούν εδώ για τη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών, ώστε να μπορούμε με κατάλληλο τρόπο να παραδώσουμε τη σκητάλη, να παραδώσουμε τους φακέλους αυτούς ε, στις, ε, στην Σουηδική Προεδρία που θα μας διαδεχτεί, διότι η συζήτηση αυτή συνδέεται στενά με την παράλληλη συζήτηση για το μέλλον των ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Για όλους τους λόγους αυτούς Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που πραγματοποιείται αυτή η διακοινοβουλευτική συνάντηση που δίνει τη δυνατότητα σε ε, βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, να ακουστεί η φωνή τους. Ε, η Τσεχική Προεδρία θα ακούσει πολύ προσεκτικά και θα υποβάλει στο Συμβούλιο, στα κράτη-μέλη που εκπροσωπούνται εκεί, μια έκθεση της συνάντησης αυτής και των όσων θα υποθούν. Κλείνοντας, ε, θα ήθελα να πω ότι οι εκδηλώσεις που θα οργανώσει η Τσεχική Προεδρία στον τομέα αυτών περιλαμβάνουν μία διάσκεψη στο τέλος του επόμενου μήνα για το μέλλον της ε, ε, πολιτικής συνοχής. Και στα τέλη του Απριλίου θα πραγματοποιηθεί άτυπη υπουργική συνάντηση. Άτυπη υπουργική διάσκεψη ε, Υπουργών ε, Περιφερειακής Πολιτικής. Οι Υπουργοί θα έχουν εκεί τη δυνατότητα να χωνεύσουν και να απαντήσουν στη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα ε, εδώ σε τούτη την αίθουσα και γενικότερα στον πολιτικό χώρο, στο δημόσιο χώρο. Στόχος είναι να ε, διοχετεύσουμε τις ιδέες που θα ακουστούν σε πολύ συγκεκριμένη ε, κατεύθυνση, καθότι είναι πολύ ευρία η συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στο Γενικό Διευθυντή του, Γενική της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζιο. Παρακαλώ. Τι και έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη ε, ευχαρίστηση και προνόμιο να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Και θα πρέπει να πω ότι το μόνο μειονέκτημα που νιώθω είναι ότι ε, πρέπει να περιοριστώ σε 10 λεπτά. Έχω τόσα πολλά να πω για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής που τα 10 λεπτά ε, μπορεί να μην μου επιτρέψουν τον ενθουσιασμό και το πάθος που έχω για την πολιτική αυτή. Δεν υπάρχει επίσημη θέση της Κομισιόν για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μέχρι στιγμής. Η θέση αυτή θα διαμορφωθεί στα πλαίσια τη συζήτηση ε, για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιμένω κάτι να δημοσιευτεί υπογραπτή μορφή ε, κατά τη διάρκεια του χρόνου. Σήμερα λοιπόν μπορώ να σας παρουσιάσω τι θέσει μου και τη δική μου κατανόηση σχετικά με την κατεύθυνση που παίρνει η συζήτηση αυτή τη στιγμή και να σα πω ποια είναι τα σημεία κλειδιά τη ε, συζήτησή μα και της ε, Γενικής Διεύθυνσης για την ε, Περιφερειακή Πολιτική. Ε, μεγάλο μέρος της συζήτησης ήδη έχει πραγματοποιηθεί. Θα θυμάστε την τέταρτη έκθεση συνοχής, τη διαβούλευση που ακολούθησε την έκθεση αυτή, την πέμπτη έκθεση προόδου για την οικονομική και κοινωνική συνοχή που παρουσίαζε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής. Ε, τα αποτέλεσμα αυτά έδειξαν σχεδόν ομοφωνία ή, εν πάση πτώση, πολύ ευρία συνένεση σχετικά με την ανάγκη να συνεχιστεί μια τέτοια πολιτική σε όλη την Ευρώπη και μετά το 2013. Είχαμε την πράσινη βίβλο για την εδαφική συνοχή και τη διαβούλευση που ακολούθησε την πράσινη βίβλο. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται τώρα και σε λίγες εβδομάδες θα ε, έχουμε μια ε, ε, εποπτική εικόνα των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης αυτής. Επίσης, στον Φαμπρίσιο Πάκα έχει αναθέσει η Επιτροπή μια μελέτη η οποία θα δημοσιευτεί τον Απρίλιο φέτος νομίζω και η Επιτροπός μου σίγουρα θα θέλει ε, να παρουσιάσει τις δικές της ε, θέσεις σε σχετική έκθεση. Η συζήτηση για το μέλλον της ε, πολιτικής συνεχής αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο ήδη αναφέρθηκε σύντομα, πρόκειται για το επίπεδο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης δύο σημαντικά θέματα προκύπτουν και τα δύο είναι ε, πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο ε, έχει να κάνει με το θέμα της αποτελεσματικότητας της πολιτικής. Πολύ δικαιολογημένο ερώτημα αυτό. Ποιος θα ήθελε να αξοδέψει 350 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια 7 ετών για μια πολιτική που δεν είναι αποτελεσματική. Κανένας δεν θα θέλει να το κάνει αυτό. Επιτρέψτε μου όμως να πω επίσης ότι έχουμε πολλά στοιχεία ήδη σήμερα που δείχνουν ότι η πολιτική αυτή είναι αποτελεσματική και στους επόμενους μήνες ε, προς το τέλος της χρονιάς. Ε, πιστεύουμε ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ε, του διαστήματος 2000-2006. Θα μπορέσουμε έτσι ίσως να προσθέσουμε επιπλέον επιχειρήματα, επιπλέον στοιχεία για το θέμα αυτό. Το δεύτερο ερώτημα, το οποίο εν μέρη μόνο συνδέεται με το πρώτο, είναι το θέμα των στόχων που θα πρέπει να θέσει η πολιτική αυτή και κύριε Πρόεδρε αναφερθήκατε σε αυτό. Ε, η ε, ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι ο λεγόμενος στόχος 2, όπως λέγοντας στο παρελθόν. Ε, από ό,τι βλέπω από τη συζήτηση αυτή, αυτή τη στιγμή μεταξύ όλων των κρατών μελών υπάρχει ευρεία συνένεση σχετικά με την συνέχιση όσον αφορά των στόχων σύγκλησης. Ε, επίσης υπάρχει ευρεία ε, συνένεση σχετικά με την προστιθέμενη αξία, ε, του τι, προσθέτει, τι αξία προσθέτει η κοινότητα στον στόχο 3 ε, για διοδοτική συνοχή. αλλά να μην ξεχνάμε ότι πραγματοποιείται συζήτηση για το στόχο 2. Δεν Νομίζω ότι και η Επίτροπος μου θα συμφωνήσει ότι εγώ προσωπικά πάντως είμαι πεπισμένος ότι για πολλούς καλούς λόγους θα χρειαστούμε επίσης πολιτική συνοχής μετά το 2013 που θα ε, ισχύει για όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, δεν υπάρχει αμφιβολία ε, το θέμα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, ε, της δημιουργίας απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον από ό,τι σήμερα. Και η παρούσα κρίση νομίζω μας θύμισε με πολύ σκληρό τρόπο πόσο απαραίτητη είναι μια τέτοια πολιτική. Ο... Ε, η επιλογή σχετικά με το στόχο 2 είναι τελικά πολιτική επιλογή και γι' αυτό είναι σημαντικό να ε, γίνει η επιλογή αυτή ε, με περιστατημένο τρόπο. Η συζήτηση όμως για την πολιτική συνοχή πείτε και σε άλλο επίπεδο. Στο επίπεδο που ασχολείται με το πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός αυτός. Πώς θα λειτουργήσει η πολιτική αυτή, τι μορφή θα έχει ο μηχανισμός. Πρόκειται για μια πολιτική για την οποία θέλουμε να ξέρουμε για το μέλλον πού χρειάζεται να βελτιωθεί η βασική ε, αρχιτεκτονική της πολιτικής μας, ε, πρέπει να πω, ε, είναι καλή κατά τη γνώμη μου. Το σύστημα συνεργασίας σε εταιρικό επίπεδο ανάμεσα στο ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι κάτι που έχει ωφελήσει όλα τα σχετικά επίπεδα όσον αφορά την, την συνεργασία. Και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα Αυτό πράγματι είναι αξία Σε πολλά σημεία όμως μπορούμε ακόμα να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Να αναφέρω τους συγκεκριμένους τομείς στους οποίους δουλεύουμε αυτή τη στιγμή για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της πολιτικής αυτής και τον ε, μηχανισμό εφαρμογής της. Καταρχήν υπάρχει το θέμα των προτεραιοτήτων. Φυσικά πρόκειται περί πολιτικής επιλογής. Και πάλι όμως ε, θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη η επιλογή. Και γι' αυτό προς το τέλος της περσινής χρονιάς δημοσιεύσαμε έκθεση με την οποία προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε μια ε, ανάλυση προοπτικής, να ε, δούμε τι αντίκτυπο θα έχει η επόμενη γενιά προγραμμάτων συνοχής, ε, γύρω στο 2020 δηλαδή και μετά το 2020. Μπορεί να πει κανεί, ότι όταν μιλάμε για το 2002 πολλά πράγματα είναι θεωρητικά φυσικά. Υπάρχουν όμως κάποιε σημαντικές τάσεις ε, τις οποίες παρατηρούμε και οι οποίες ε, το πιθανότερο είναι θα συνεχίσουν ε, να υπάρχουν. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν αυτές οι τάσεις τι επίπτωση θα έχουν στην κατάσταση τη περιφέρεια σε όλη την Ευρώπη. Σκεφτείτε την αλλαγή του κλίματος. Σκεφτείτε την ε, ε, παγκοσμιοποίηση, σκεφτείτε τις δημογραφικές εξελίξεις, σκεφτείτε ε, το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, σκεφτείτε τα αυξανόμενα προβλήματα που έχουμε όσον αφορά την κοινωνική πόλωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αναλύσουμε στην έκθεσή μας αυτή τη, μέχρι στιγμής έχουμε επικεντρωθεί ε, στους, στις πέντε οικονομικές πτυχές. Ε, συνεχίζουμε όμως τις εργασίες μας πάνω στις κοινωνικές πτυχές ε, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση. Και θα θέλαμε να καταλήξουμε σε μια επισκόπηση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει η κοινωνία μας το 2020 και την επίπτωση των προβλημάτων αυτών στο περιφερειακό επίπεδο. Παρουσιάσαμε λοιπόν ε, αυτή τη δημοσίευση διότι θέλουμε να ε, προκαλέσουμε ε, τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη να κάνουν παρόμοιες αναλύσεις ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα προβλήματα αυτά και στο τέλος να έχουμε μια ευρωπαϊκή επισκόπηση όπου η κάθε περιφέρεια θα είναι ένα παραθυράκι που μπορούμε ε, να ανοίξουμε και να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές για τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Είναι φιλόδοξο το σχέδιο αυτό, ε, θέλουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας ε, σε αυτό όμως. Και υπάρχει άλλος ένας ε, τομέας όπου θέλουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Θέλουμε να μην βλέπουμε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση απομονωμένη. Το τι θα συμβεί τα επόμενα 15-20 χρόνια γύρω από την Ευρώπη, το τι θα ε, πραγματοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και ποιες θα είναι οι συνέπειες ε, για την Ευρώπη. Ένα παράδειγμα. Φανταστείτε μια σειρά δημοσίευσεων ε, για την, ε, για την αλλαγή του κλίματος που να λέει ότι τα επόμενα 30-40 χρόνια ε, θα έχουμε μισό εκατομμύριο μετανάστες στον κόσμο λόγω της αλλαγής του κλίματος. Ποιες θα είναι οι συνέπειες της μετανάστευσης αυτής για την Ευρώπη και τι μπορούμε να κάνουμε για να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Πρόκειται για μια σειρά ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν. Και ε, κύριε Πρόεδρε, βλέπω ήδη σήμερα στη συζήτηση αυτή ότι η παγκοσμιοποίηση θα παραμείνει κεντρικό θέμα, η αλλαγή του κλίματος ε, θα γίνει σημαντικό θέμα και σε μια σειρά περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε, θα είναι και οι δημογραφικές αλλαγές μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν, έχει, ε, δεν έχουν συνειδητοποιήσει όλοι ακόμα. Ε, και υπάρχει και ένα άλλο θέμα πάνω στο οποίο εργαζόμαστε, την ανάπτυξη των αστικών και υπαίθριων περιοχών και τον σχετισμό μεταξύ τους τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της πολιτικής μας για να φανεί η πτυχή ε, αυτή πιο πολύ στο μέλλον. Ε, θυμάμαι ότι αυτό το θέμα έχει συζητηθεί και στην Επιτροπή σας. Πρέπει να ξεπεράσουμε την παλιά ξεπερασμένη διχοτομία ανάμεσα στην ανάπτυξη των υπαίθριων περιοχών από τη μία και την ανάπτυξη των αστικών περιοχών από την άλλη μεριά. Στενά με αυτά συνδέεται ένα θέμα ε, το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε περισσότερο. Πρόκειται για, το, για τις ε, πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης. Ε, είχαμε στο παρελθόν κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως ήταν το Leader ή το Urban που βασίζονταν σε ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη. Και Έχω λίγο την εντύπωση ότι με την απλοποίηση ε, στον τομέα της αστικής ανάπτυξης που παρακολουθώ εγώ πιο στενά χάνουμε αυτή την ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση και θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό διότι φοβάμαι ότι θα χάσουμε κάτι ε, στην πολιτική μας που έχει μεγάλη αξία. Και ένα ακόμα θέμα ένα άλλο θέμα σημαντικό για μας είναι η εδαφική συνεργασία, η διασυνοριακή συνεργασία, η ε, συνεργασία μεταξύ των χωρών και η διαπεριφερειακή συνεργασία. Πιστεύω ότι υπάρχει συνένεση σε όλη την Ευρώπη ότι η εδαφική συνεργασία ε, μπορεί να έχει το ρόλο του τρίτου πυλώνα της ε, πολιτικής συνεχής. Ε, υπάρχει ακόμα πολύ δυναμικό ανάπτυξη στον τομέα αυτών και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό αυτό. Πρόκειται για έναν πυλώνα όπου η ευρωπαϊκή προοπτική, η υπερεθνική προοπτική, η προστιθέμενη αξία από το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι προφανής είχαμε ενδιαφέρουσες εξελίσεις τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες. Ε, βλέπουμε νέο ενδιαφέρον στο τομέα της εδαφικής συνεργασίας που συνδέεται ιδιαίτερα με την ε, διασυνοριακή συνεργασία. Σκεφτείτε τη στρατηγική της Βαλτικής. Μια σειρά από χώρες και περιφέρειες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα προσπαθούν να συνεργαστούν ώστε να λύσουν από κοινού τα προβλήματα αυτά και ζητούν από την Επιτροπή να τους βοηθήσει να διαμορφώσουν μια στρατηγική, ένα σχέδιο δράσης, ένα σύστημα το οποίο να λειτουργεί και το οποίο να μπορέσει να ε, οργανώσει αυτή τη συνεργασία. Ε, άκουσα ότι υπάρχει παρόμοια ενδιαφέρον ε, στην περιοχή του Δούναβη για να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διακρατικές μορφές συνεργασίες που μπορούν να παίξουν πιο σημαντικό ρόλο στο μέλλον και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε το 2012 να σας παρουσιάσουμε ένα πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει αρκετή ευελιξία ε, ώστε να μπορούν να, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον συνεργασίας και αυτό σε αντίθεση με τις πιο κλασικές μορφές διακρατικής συνεργασίας που παραμένουν σημαντικές. Γρήγορα θα αναφερθώ σε κάποιους άλλους ε, τομείς να αναφερθώ ε, στο ότι πρέπει να κοιτάξουμε καλύτερα ε, την καλύτερη συνεργα... τον καλύτερο συντονισμό με άλλες πολιτικές, άλλες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. Πώς μπορούμε να τις οργανώσουμε αυτές στο μέλλον. θα θέλαμε σε συνεργασία μαζί σας εξετάσουμε το ερώτημα πώς μπορούμε περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν να αντί για επιδοτήσεις να χρησιμοποιήσουμε ε, άλλα ε, ε, χρηματοδοτικά μέσα, δάνεια, κεφάλαια επιχειρηματικά, πράγματα που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι τόσο σημαντικές για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της καινοτομίας. Πρόκειται λοιπόν για έναν τομέα στον οποίο θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερη προσοχή. Σκεφτείτε το πλεονέκτημα. Αν χρησιμοποιήσουμε περισσότερα τέτοια χρηματοδοτικά μέσα, αυτό σημαίνει ότι ε, τα χρήματα που επενδύουμε ε, έρχονται πίσω, ε, μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Οι δημόσιοι πόροι δηλαδή μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για παρόμοιους στόχους. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και εξετάζουμε αυτό το Τζέρεμι, Τζέσικα, κοιτάμε τα ανακυκλούμενα κεφάλαια και είναι κάτι το οποίο θα προσέξουμε πολύ περισσότερο στο μέλλον. Και τέλος έχουμε τα ερωτήματα που πάντα ανακύπτουν και έχουν να κάνουν με την απλοποίηση, λιγότερη γραφειοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι παίρνουμε απολύτως στα σοβαρά το ερώτημα αυτό. Δεν είναι απλά κάτι που χρησιμοποιούμε στις ε, κυριακάτικες ομιλίες μας. Συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για να εξετάσουμε προσεκτικά τους, ε, τις παρούσες διατάξεις ε, και τα μελλοντικά προγράμματα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να απλοποιήσουμε τη ζωή για τα κράτη-μέλη, αλλά και, και ακόμα περισσότερο ίσως, για τους ε, τελικούς ε, δικαιούχους. Ε, ήδη έχουμε παρουσιάσει κάποιες προτάσεις απλοποίησης. Αργότερα θα υποβάλουμε επιπλέον προτάσεις και το πρώτο πράγμα που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι ο κανονισμός της ε, Κομισιόν οι κανονισμοί της Κομισιόν, οι διατάξεις της Κομισιόν όπου μπορεί να ε, πραγματοποιηθεί ε, πολλή ε, δουλειά απλοποίησης κατά τη γνώμη μας. Όταν όμως κοιτάμε το χρόνο μετά το 2013, από την αρχή, από αυτή τη στιγμή και μπρος δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε περιτές περιπλοκές που θα πρέπει να διορθωθούν εκ των υστέρων. Έτσι κάποιες πινελιές εξπρεσιονιστικές σας έδωσα κύριε Πρόεδρε για να σας δώσω μια επισκόπηση ε, της δουλειάς μας. Περιμένω όμως με πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τις προτάσεις της παρούσας συνέλευσης ε, και ε, θα κρατήσω σημειώσεις για τη μελλοντική μας δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γενικέ. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι αν γίνει δεκτή η σύνθηκη της Σαββόνα και τεθεί σε ισχύ, θα υπάρξει ειδική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών κοινοβουλίων. Είναι η περίφημη κίτρινη κάρτα και η δυνατότητα που έχουν οι βουλευτές, οι εθνικοί βουλευτές να επηρεάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γι' αυτό είναι και τόσο σημαντική η συνεργασία μας και μάλιστα πάρα πολύ στενή συνεργασία. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα για τη συζήτηση. Α, όχι, έχουμε και άλλες εισαγωγικές ομιλίες. Πριν ανοίξω τη συζήτηση, εγώ φταίω, έκανα λάθος. Θα ακούσουμε δύο διαφορετικές πρόπτικες. Έχουμε την τσεχική πρόπτικη, τον κύριο Μπάρεκ από τη τσεχική Γερουσία, που είναι η σημερινή προεδρία. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε την επόμενη προεδρία, τη Σουηδική, που εκπροσωπείται εδώ από το Σουηδικό Κοινοβούλιο και η συζήτηση ακολουθεί. Ε, κύριε Μπάρεκ, έχετε μέσα στο λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Γενικέ, Διευθυντά, αγαπητοί συνάδελφοι. Για μένα αποτελεί μεγάλη τιμή η ευκαιρία που έχω σήμερα να σα απευθύνω το λόγο για να αρχίσουμε μια συζήτηση για την πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα δεν είμαι ο μόνος εγώ που θεωρώ ότι η πολιτική αυτή είναι σημαντική όχι μόνο για τα ποσά που επενδύονται, θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα είναι μια πολιτική που διακρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με ε, άλλες ε, διακρατικές οργανώσεις. Εκταμιεύονται πόροι από τα διαρθωτικά ταμεία προς τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες και αυτές είναι πολιτικές της Ένωσης που επιτρέπουν να δίνουμε ε, θετική εικόνα για την Ένωση την κοινή γνώμη, με την ευρία έννοια. Βεβαίως, ε, κυρίω εγώ περιμένω να ακούσω τη συζήτηση και τις απόψεις που θα ανταλλάξουμε, καθώ και τι εθνικές εμπειρίες για το πώ μπορούμε ακόμα στο μέλλον να βελτιώσουμε τα πράγματα. Πολύ σύντομα θα ήθελα να ε, σας παρουσιάσω τις δραστηριότητες της τσεχικής γερουσίας από πλευρά συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται στο μέλλον, ποιο θα είναι το κέντρο ενδιαφέρον και πώς σκεφτόμαστε να έχει μελλοντικά η πολιτική συνοχής. Θα ήθελα να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι ε, σε αντίθεση ε, με άλλα κοινοβούλια ε, που έχουν δύο βουλευτικά σώματα, η δική μας γερουσία δεν εκπροσωπεί τις περιφέρειες. Έχει 81 γερουσιαστές που εκλέγονται από όλη τη χώρα, από εκλογικές περιφέρειες ε, καλύπτοντας όμως το σύνολο της τσεχικής δημοκρατίας. Δεν είμαστε εκπρόσωποι περιφερειών στην τσεχική Ιερουσία. Σε άλλες χώρες είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, για τη Δημόσια Διοίκηση, την Περιφερειακή Ανάπτυξη και το Περιβάλλον, της οποίας προεδρεύω, έκανε ακρόαση με τεχνικά στη συνέχεια σε σεμινάρια που είχαν αφιερωθεί στην δυνατότητα απορρόφησης των χρηματικών πόρων από τα διαρθωτικά ταμεία, από την Τσεχία. Ε, συμμετέχει στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ή μάλλον του, του θετικό ελέγχου και παίζει σημαντικό ρόλο η γερουσία σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή ε, στον καθορισμό των πολιτικών της κυβέρνησης και στην τοποθέτηση της κυβέρνησης για τα συγκεκριμένα νομοσχέδια. Το τελευταίο κείμενο που μας απασχόλησε είναι η πράσινη βίβλος για την κοινωνική συνοχή. Και μάλιστα το συζητάμε ακόμα. Ε, ποιο είναι για μας το σημαντικότερο ή τα βασικότερα στοιχεία και πώς φανταζόμαστε στο μέλλον την πολιτική συνοχής. Ε, μια βασική αρχή που θα πρέπει να διατηρηθεί είναι η ιδέα που έχουμε για την αλληλεγγύη. Η υποστήριξη στα κράτη-μέλη και στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες για να μειωθούν οι ανισότητες που έχουμε στο επίπεδο ανάπτυξής τους. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της υποστήριξης θα πρέπει εδώ να συμπεριλάβουμε τις αντιδράσεις στις νέες προκλήσεις που είναι η οικονομική μεταρρύθμιση, η δημογραφική γύρανση και η κλιματική υπερθέρμανση όλα αυτά έχουν επιπτώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις περιφέρειες και κινδυνεύουν να οξύνουν ακόμα περισσότερο τις ήδη υπάρχουσε διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Θα ήθελα εδώ να θυμίσω μία από τις λειτουργίες της πολιτικής συνοχής που δεν την αναφέρουμε συχνά. Η κοινωνική μάλλον η, πολιτική συνοχή παίζει και ένα ρόλο σταθεροποιητικό ε, γιατί αναδιανέμει πόρους ε, στις χώρες και τις περιφέρειες που είναι λιγότερο ευνοημένες και έτσι έχουμε τελικά και οικονομική σύγκληση. Η οικονομική σύγκληση είναι απαραίτητη για τις ε, χώρες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, μεν, αλλά είναι και επιθυμητή για τις χώρες που πρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα φιλοδοξούν να ε, υιοθετήσουν το ενιαίο νόμισμα. Και ιδιαίτερα στη σημερινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που διανύουμε θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας αυτά. Γι' αυτό καλωσορίζουμε τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της κρίσης, διότι ακριβώς εκεί εστιάζονται στη χρήση ε, των ε, εργαλείων αυτών για να ενισχυθεί η οικονομία και να λυθεί η οικονομική κρίση. Η πολιτική συνοχή λοιπόν συνεισφέρει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Λισαβόνας. Ωστόσο, η πολιτική συνοχή δεν θα έπρεπε να περιορίζεται στην απλή χρήση των εργαλείων προς την κατεύθυνση αυτή. Για τη στρατηγική της Λισαβόνας τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά με ε, τα ε, εθνικά σχέδια και τα μεταρρυθμιστικά. Αυτή τη στιγμή μιλούμε περισσότερο για την τρίτη διάσταση της πολιτικής συνοχής, τη διάσταση, τη λεγόμενη εδαφική ε, αποτέλεσμα και απόδειξη είναι η πράσινη βίβλος που το φθινόπωρο κυκλοφόρησε, εντάσσεται σε αυτή την πολιτική συνοχή. Όπως σας είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου, Όλα αυτά τα εξετάζει η αρμόδια επιτροπή μας στη Γερουσία, αλλά θέλω να σας πω ότι θα υποστηρίξουμε την τσεχική κυβέρνηση γιατί οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών δεν είναι μόνο ε, γεωγραφικού χαρακτήρα. Ε, θα πρέπει να δούμε το ανθρώπινο δυναμικό, την πρόσβαση, τις τεχνολογίες, τις υπηρεσίες. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη γεωγραφική ή τη φυσική ή την εδαφολογική κατάσταση. Για μας η, κοινωνική, η εδαφική συνοχή συγγνώμη, θα πρέπει να συμβαδίζει με την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και με χαρά περιμένω να ακούσω τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Βάιμπουλ που είναι από την Επιτροπή ε, Βιομηχανίας και Εμπορίου της Σουηδικής Βουλής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να... Σας ε, ε, πω ότι η συζήτηση για την πολιτική συνοχή μετά το 2003 θα βασιστεί στον προπολογισμό που θα της δοθεί μέχρι το 2003 προορίζεται για τα κράτη-μέλη τα οποία ε, είναι φτωχότερα τόσο όσον το επίπεδο ζωής όσο και το επίπεδο εσόδων. Να, στόχος είναι να συμπληρωθούν κάποιες φυστάμενες ελλείψεις. Άρα λοιπόν αυτές οι περιοχές με υστέρηση θα μπορούν έτσι να λάβουν κάποια βοήθεια. Είναι η στρατηγική αυτή πτυχή της συνοχής που επιτρέπει την ε, αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων πόρων. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να συμβάλλουν στην μείωση των διαφορών και να αυξήσουν την ανταγωνιστική δυνατότητα των περιφερειών που ορισμένες από αυτές είναι ιδιαίτερα Βέβαια. Ε, Καθυστερημένε Υπάρχουν περιφέρειες που έχουν το δυναμικό και που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ε, τους πόρους αυτούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζουμε πως αυτή είναι, αυτό είναι το θεμέλιο της πολιτικής συνοχής και ε, καθιερώνεται και από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ελπίζουμε η συνθήκη της Λισαβόνας να μπορέσει να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και να δώσει τις βάσεις, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ε, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο χώρο για να αναπτυχθούμε. Τα στην ε, Σουηδία αφορούν ε, την, ε, ε, τον ανεφοδιασμό σε ενέργεια, την, καινα, την καινοτομία και γι' αυτό και θα πρέπει η πολιτική συνοχή να βοηθήσει τις περιοχές της Ευρώπης να εξυγχρονιστούν, να ασχοληθούν με την καινοτομία και με τη γνώση για να μπορέσουν να απαντήσουν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να βοηθήσει τις περιφερειακές οικονομίες ώστε να βρουν τη θέση τους στις παγκόσμιες αγορές. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία και ποια είναι τα αδύναμα σημεία και να χρησιμοποιηθούν τα δυνατά σημεία για την ανάπτυξη. Γι' αυτό και θα πρέπει να αναπτυχθούν και νέες ε, ε, δεξιότητες. Πολύ συχνά τα προγράμματα δεν υλοποιούνται, δεν συγκεκριμενοποιούνται. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσαμε να δώσουμε οικονομική στήριξη. Βεβαίω μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά που υπάρχουν. Υπάρχουν και κάποια μεγάλα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν από κοινού να χρηματοδοτηθούν και που θα μπορούσαν να έχουν εφέ ε, χιονοστιβάδας για την ανάπτυξη και που θα μπορούσαν επίσης να έχουν ε, ε, μακροπρόθεσμους στόχους με μεγάλη προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τομείς όπως η ενέργεια, οι τεχνολογίες που συνδέονται με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και ένα σωρό άλλοι τομείς εχμής όπου μπορούμε πραγματικά να ε, έχουμε ε, αριστεία. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και να αντιποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Για κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να κάνουμε μια σωστή ανάλυση, αλλά και να αναλάβουμε η πολιτική της ευθύνης μας με πνεύμα δημιουργικό. Εμείς έχουμε ευθύνη, φέρουμε ευθύνη, ε, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν τομείς που έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα, κλίμα, ενέργεια, περιβάλλον θα μπορούσαν αυτά να θεωρηθούν ένα σύνολο προτεραιότητας και επίσης ε, στο διασυνοριακό επίπεδο σίγουρα είναι πιο κέρια. Ε, και κάθε περιφέρεια έχει βέβαια τις ιδιαιτερότητές της. Ε, εμείς έχουμε την στρατηγική του Όστερσεβ, δηλαδή την περιοχή που πάει από την Κοπενχάγη μέχρι το Μάλμο και θεωρούμε όλη αυτή την περιοχή ως μία περιφέρεια και θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες δυνατότητες και να εξελιχθούμε περισσότερο δημιουργώντας έτσι θέσεις απασχόλησης, δυνατότητες απασχόλησης από τη στιγμή που έχουμε ε, αυτήν την προ... την στρατηγική αυτή του Έστερσουρ, όπω σα είπαμε, από την Κοπεχάγη μέχρι το, που είναι στη Δανία μέχρι το Μάλμε στη Σουηδία. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει πηγή έμπνευση για άλλες περιφέρειες. Βέβαια τα προγράμματά μας δεν περιορίζονται μόνο σε αυτή την περιφέρεια. Υπάρχει συνεργασία και με άλλες χώρες της ε, Βαλτικής θάλασσας. Η στρατηγική αυτή έχει να κάνει με 6 εκατομμύρια ανθρώπους. Ε, επιτρέπει μια εξέλιξη και ε, σε διάφορους τομείς, δηλαδή η διασυνοριακή ανάπτυξη υποδομών, μεταφορές, αυτό αποτέλεσε την ε, ε, τη χιονοστιβάδα που επέτρεψε αυτήν την ε, ανάπτυξη. Μία περιφέρεια μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη που και να τραβήξει, να προσελκύσει και άλλες περιφέρειες που βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση. Αυτό περιμένουν οι πολίτες μας σε κάθε περιφέρεια, στα κράτη-μέλη, να μπορέσουν να συνεργαστούν, ώστε να έχουν αυτό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, διαφορετικά όχι. Αυτό σημαίνει η συνεργασία σε διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να προσπαθήσουμε, όπως είπαμε, να περιοριστούμε πάνω κάτω στα τρία λεπτά. Ο κύριος Κλάους Σέχ από την Bundesrat της Γερμανίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω. Για σηκώστε κανένα χέρι να σας δούμε που κάθεστε. Οι ομιλητές, όχι όλοι. Ωραία, ευχαριστώ και πάλι για τη δυνατότητα που μου δίδετε. Μιλώ ως εκπρόσωπος της Άνω Βουλής Γερμανίας, Bundesrat, που εκπροσωπούνται τα ομόσπονδα κρατήδια. Και θέλω ευθύ εξ αρχής να σας πω ότι ζω και εργάζομαι σε ένα από τα κράτη-μέλη που είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία, στην πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Και πραγματικά θέλω να τονίσω ότι και βλέπουμε και ζούμε καθημερινά τις θετικέ επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί και στην πολιτική απασχόληση και στην προώθηση και πανένταξη των μακροχρόνιων ε, ανέργων στην αγορά εργασίας, αλλά αυτό φαίνεται και από τη βελτίωση των ευκαιριών των γυναικών στην αγορά εργασίας και η απαραίτητη και χρήσιμη υποστήριξη εγκατάστασης ε, εταιριών, βιοτεχνών ε, και βιομηχανιών. Με την ε, μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής στη Γερμανία γίνονται βαθιές μεταρρυθμίσεις. Το μέλλον της διαρθρωτικής πολιτικής για μας σημαίνει συνέχεια των σημερινών κατευθυντηρίων γραμμών. Οι ε, ισχυρές πτυχές θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο και οι αδυναμίες να καλυφθούν. Άκουσα το Γενικό Διευθυντή κύριο Dirk Άνερ και με χαρά ε, διαπιστώνω και ακούω αυτό που λέτε ότι στη διοίκηση θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Στη διοικητική μηχανή απασχολούνται πολλοί υπάλληλοι για να διεκπαιρώνουν αυτές τις διαδικασίες και θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε πολύ καλύτερα αλλού. Βασικός στόχος της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να είναι η άρση των οικονομικών και των κοινωνικών διαφορών. Αυτός ο στόχος είναι σημαντικός πυλώνας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να ενισχύει τις περιφέρειες που έχουν υστέρηση ανάπτυξης και αυτό να το έχει στο μυαλό της και στο μέλλον. Θα πρέπει κυρίως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στην περιφέρεια και η απασχόληση ε, και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Από τη δική μας σκοπιά δεν θα πρέπει να υπάρχει απότομη διακοπή της χρηματοδότησης. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που μετά τις μεταβατικές διατάξεις δεν θα είναι στην ανώτατη κατηγορία στήριξης. Ε, αυτό θα διακυβεύσει τις επιτυχίες που είχαμε μέχρι τώρα, αν απότομα επαναλαμβάνω σταματήσει χρηματοδότηση. Γι' αυτό εμείς ζητούμε βεβαίως να υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι, αλλά σωστές και κατάλληλες για τις περιφέρειες που βγαίνουν από την πρώτη στήριξη. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει συμμεταχείριση στην Ευρώπη και προφανώς υπάρχουν πολλά σημεία για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ε, της αποδοτικότητας ευρωπαϊκής πολιτικής ε, συνοχής, ιδιαίτερα στη σημερινή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Ιδιαίτερα τότε βλέπουμε ότι η απλούστευση της εκταμίευσης των πόρων είναι πολύ σημαντική κατεύθυνση και θα πρέπει να ακολουθηθεί. Η έκθεση συνοχής, η τέταρτη, μιλάει ε, για ε, πολλές νέες προκλήσεις και ακούστηκε ιδιαίτερα το θέμα των κλιματικών αλλαγών και της προμήθειας ενέργειας. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε οι νέες προκλήσεις να απαντηθούν με νέες πολιτικές πρωτοβουλίες και η πολιτική συνοχή να μην υπερφορτωθεί πολύ με νέους στόχους και στην επιλογή των ε, δικτών για τις ε, πιο φτωχές περιφέρειες θα πρέπει να είναι και το ΑΕΠ κατά κεφαλή και αυτός είναι ο μόνος δείκτης ο οποίος είναι επιστημονικά αναγνωρισμένος και σχετικά εύκολος να μετρηθεί. Επίσης θέλουμε μια σύγχρονη πολιτική που να μπορεί να τη χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος όλων, αλλά ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι κοινότητες θα πρέπει να έχουν και κάποιο περιθώριο λιγμών και κινήσεων ε, για αποκεντρωμένη διαχείριση. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκασπάρ Τζίτσι από τη Βουλή της Ιταλίας στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Ο κύριος Τζούντιτσε Γκασπάρ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συζήτηση για την πολιτική συνοχή είναι μια σημαντική δοκιμασία αποφασιστική για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί η πολιτική συνοχή θα εξαρτηθεί η ίδια ιδέα της Ευρώπης. Η συνοχή είναι μια από τις βασικές αξίες της ευρωπαϊκής ε, οικοδόμησης ως έκφραση ελεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη και είναι ένας ε, όρος εκ των όνων κάνευ για την ανάπτυξη της, της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ανταγωνιστική οικονομία, αλλά αυτό εις βάρος της εσωτερικής συνοχής και με τη διατήρηση των αρχών της αλληλεγγύης, την προστασία των, των δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, που είναι μια από τις πιο ψηλές αξίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωση Ενώπιον τη ε, διεθνού χρηματοπιστωτική κρίσης, η πολιτική συνοχή κατέστη ω ένα διαμφισβήτητο μέσο, γιατί η κρίση ε, προκαλεί εντατικά ε, εντυνόμενα προβλήματα σε διάφορες περιφέρειες. Το κλείσιμο πολλών βιομηχανιών αλλά και η απώλεια πολλών θέσεων απασχόλειας είναι πολύ ε, πιο σοβαρές στις ε, περιοχές με υστέρησης. Η διεύρυνση που έγινε και η κεντρική ρύθμιση της πολιτικής συνοχής αποτέλεσαν το βασικό εργαλείο για την εγγύηση της ένταξης και της ολοκλήρωσης των νέων κρατών μελών. Δεν αμφισβητείται πλέον ο πρωταρχικός ρόλος της πολιτικής συνοχής ε, σε σχέση με τις υπόλοιπες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αποδεκτή η πρόταση για την επανεθνικοποίηση της, περιφερειακής, της πολιτικής συνοχής. Δεν μπορεί να φανταστούμε να, ξα... να, να αποκλειστούν τελείως οι παλιές περιοχές των παλιών κρατών μελών από τα ταμεία συνοχής γιατί τα αποτελέσματα είναι προφανή. Η Ιταλία και πολλά άλλα κράτη-μέλη το δέχτηκαν σε συνέπεια με την αρχή της ε, αλληλεγγύης, δέχτηκαν δηλαδή πολλές μειώσεις ε, για τις δικές τους περιφέρειες για την περίοδο 2007 και μέχρι 2013 λόγω της διεύρυνσης στα νέα κράτη-μέλη. Η επόμενη προγραμματική περίοδος μπορεί να βασιστεί σε, σε διαφορετικά θεμέλια λόγω των σημαντικών προόδων που, ε, που επέτυχαν τα νέα κράτη-μέλη. Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε σταθεροί σε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, η πολιτική συνοχή είναι η περιφερειακή πολιτική. Η αναφορά η εδαφική δεν μπορεί παρά να είναι η περιφέρεια, γιατί διαφορετικά θα εκφυλιστεί η ίδια η πολιτική συνοχή. Το λέει και η συνθήκη της Λισαβόνας όπου εισάγεται σαφώς η εδαφική ε, ε, ε, διάσταση της περιφερειακής πολιτικής. Δεύτερον, η πολιτική είναι και πρέπει να παραμείνει μια πολιτική στήριξη στην απασχόληση και στην ανάπτυξη των λόγων περιφερειών. Και γι' αυτό θα πρέπει να αποφευθεί οποιοδήποτε πειρασμός λισαβονοποίησης για την ένταξη διαφόρων άλλων στόχων, για τους οποίους θα πρέπει να προσφύγουμε σε άλλα πολιτικά και οικονομικά μέσα. Τρίτο σημείο, η πολιτική συνοχή θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί πόρους ε, όπως αυτοί που προβλέπονται για, από το σημερινό ισχύον πλαίσιο. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τη σημαντική συμβολή των ε, πόρων και των μηχανισμών ε, χορήγησής τους. Θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να μπορέσει να, να, να περιορίσει και να στοχεύσει τους πόρους του σε συγκεκριμένους στόχους με ψηλή προστιθέμενη αξία ώστε να έχει αποτελέσματα για τις συγκεκριμένες περιοχές και κυρίως ε, τις υποδομές. Δηλαδή θα πρέπει όπως έλεγε ο προηγούμενος ομιλητής να απλοποιηθεί η διαδικασία και η μέθοδος προγραμματισμού και διαχείρισης ωστόσο με εγγύηση της ε, αυστηρότητας των μηχανισμών δαπανών και ελέγχου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Βουλευτά και σας ευχαριστώ για την πειθαρχία που δείξατε. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπέρεντ που είναι μέλος του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι καταρχάς που όλοι εδώ συμφωνούμε για το στόχο μας, αν μη τι άλλο, ότι μια ουσιαστική και δυναμική πολιτική συνοχή θα πρέπει να συνεχίζει να ισχύει στην Ένωση μετά το 2013. Και δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά τώρα σε αυτή την προγραμματική περίοδο έχουμε τόσα πολλά χρήματα, 42 44,2%. Χρόνια ολόκληρα ήταν πρώτη γεωργία, τώρα έχει περάσει συνοχή πρώτη και αυτό δεν είναι τυχαίο και σημαίνει κάτι. Και ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Πολιτικής θέλω να πω ότι και η δική μας Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχει μεγάλη συμμετοχή ακριβώς στο ότι καταφέραμε να βάλουμε το κέντρο βάρου στην πολιτική συνοχή για την παρούσα προγραμματική περίοδο αλλά και για την επόμενη. Και όπως βλέπουμε στην τέταρτη έκθεση για τη συνοχή που έφυγε από αυτή την Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι περιφερειακές και διαπεριφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο έντονες από ό,τι στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, στις περιφέρειες μεταξύ τους. Ταυτόχρονα σχεδόν μπήκαν 14 νέα κράτη-μέλη και αυτό οδήγησε σε κάποιες ε, ε, ίσως ε, αδυναμίες ε, ή διαφορές στις στατιστικές. Παρόλα αυτά παραμένουν μεγάλες οι διαφορές. Είτε πρόκειται για την τεχνολογία, για τις υποδομές, για τις συνδέσεις, για την ποιότητα ζωής κτλ. Έχετε δίκιο κύριε Γενικέ, έχουμε και άλλες προκλήσεις τώρα που μας περιμένουν από το 2013. Περισσότερο από ποτέ. Να δούμε τι θα γίνει τα, τελευταία, τα επόμενα χρόνια και πόσο θα αυξηθούν αυτές ο πληθυσμός ε, συγκεντρώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, μεγάλη αστιφιλία. Πρόβλημα. Γιατί έχουμε ε, χρόνια υπερφόρτωση ε, του συγκοινωνιακού συστήματος και έχουμε προβλήματα στις πόλεις. Επίσης, οι δημογραφικές αλλαγές που έχουμε υπεργύρανση τελικά του πληθυσμού. Διάφορα μεταναστευτικά ρεύματα. Κάποιος το ανέφερε. Επίσης η παγκοσμιοποίηση και η μεγαλύτερη ζήτηση γεωργικών προϊόντων, οι κλιματικές αλλαγές. Είναι και πιο ευάλωτες μερικές περιφέρειες έτσι σε θεομηνίες. Οι τιμές της ενέργειας που αυξάνουν. Όλα αυτά είναι προκλήσεις που θα τις βρούμε μπροστά μας την επόμενη περίοδο. Ακριβώς στην πολιτική συνοχή και όχι μόνο. Και σε αυτές τις νέες προκλήσεις πραγματικά παίρνει νέα διάσταση η ανάπτυξη της περιφέρειας για να διατηρήσουμε τα ε, μέτρα της ε, πολιτικής αυτής των διορθωτικών ταμείων οπωσδήποτε μετά το 2013 και να τα επεκτείνουμε. Και ένα τελευταίο να πω. Ε, το κέντρο βάρους δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά στα νέα κράτη-μέλη, γιατί οι προκλήσεις είναι σημαντικές για την Ευρώπη των 15 και όχι των 27. Και αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη προσέγγιση από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Για να μην μακρηγορώ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, όλες οι προτάσεις που στο μέλλον θα θέλουν να ε, ενισχύσουν μόνο το στόχο 1 και να αφήσουν στην άκρη το στόχο 2, θα πρέπει να μας βρουν αντιμέτωπους ε, απέναντί τους. Και οποιαδήποτε επίσης απόπειρα επανεθνικοποίησης της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν προσέξατε ότι στην ευρωπαϊκή συζήτηση χρησιμοποιούμε ακόμα τον όρο νέα κράτη-μέλη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση του ποιο είναι νέο, ποιο είναι παλιό και πόσο καιρό ακόμα η Πολωνία θα είναι νέο κράτος μέλος. Θα το δούμε. Θα παρακαλούσα ένα μέλος ε, κοινοβουλίου από ε, νέο κράτος μέλος να πάρει το λόγο. Κυρία Ντανούτα Γιασλοφιέσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής ήταν γενική η συζήτηση. Θα ήθελα να επικεντρωθώ ε, τις ε, εμπειρίες μας ε, ήθελα να πω πόσο χρόνο παίρνει το να αλλάξουμε τον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή ε, στη χώρα μου γίνεται μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης που σκοπό έχει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των πολιτών μας στην αγορά εργασίας, να βελτιώσει την κινητικότητα στην αγορά εργασίας, όχι μόνο από την Πολωνία αλλά και εντός της Πολωνίας. Ο Διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση ε, Ρέτζιο μίλησε για την ε, σημασία των τοπικών πρωτοβουλειών και θέλουμε να τι ενισχύσουμε αυτέ, το οποίο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τεχνική και κοινωνική υποδομή. Αυτό στοιχίζει όσο και ε, ένα νέο αυτοκινητόδρομο. και εάν η Ευρώπη θέλει να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, τότε η μελλοντική τη περιφερειακή πολιτική, θα πρέπει, η πολιτική συνοχή θα πρέπει να στηρίζεται στι κοινωνικέ εξελίξει και στο ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί το Νομπέλ Γιατρικής, ε, ε, Φυσικής ε, και, και λοιπά πάντα πάνε στους Αμερικάνους. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Υπό τις παρούσες συνθήκες της παγκόσμιας κρίσης θα πρέπει να κάνουμε τους πολίτες μας καλύτερους και πιο καλά εκπαιδευμένους. Ευχαριστώ πολύ Δίνω το λόγο στον κύριο Ιουτζένιο Νασάρα από την Ισπανία. Έχετε το λόγο. Eh. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ εγώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να διοργανώσει αυτή τη συζήτηση, διότι μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ επίκαιρη και σκόπιμη. Θα ήθελα να σας διαβιβάσω το εξής. Στην Ισπανία, στη Βουλή, την Ισπανική, όντως ανησυχούμε για το μέλλον της πολιτικής ε, κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα μετά από τις συνέπειες της κρίσης, της μεγάλης οικονομικής κρίσης που σήμερα ζούμε. Και δεν μπορούμε βέβαια να αρνηθούμε ότι Υπάρχουμε, έχουν ανισχυτικά συμπτώματα εμφανιστεί προστατευτισμού που έρχονται σε αντίθεση με τις πολιτικές συνοχής. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα πιο ασυνάρτητο από το να κάνεις προστατευτισμό στην οικονομία διατηρώντας πολιτικές συνοχής. Είναι αντιφατικά αυτά τα στοιχεία μεταξύ τους. Το πρώτο λοιπόν που θα ήθελα να σας πω είναι τουλάχιστον οι Ισπανοί βουλευτές, αυτό πιστεύουμε, ε, η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να μείνει σημαντικός παράγον στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Ιδέα δεύτερη. Βλέπουμε από την κρίση επίσης ότι η νέα στρατηγική και η πολιτική συνοχή θα πρέπει να συνδέονται όλο και περισσότερο με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πνεύμα της Αττικής Λισαβόνας που εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες να οικοδομήσουμε μια μεγάλη ε, ε, κοινωνική και οικονομική δυναμική και αυτά όλα να είναι μοχλή για να συνεισφέρουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ιδέα τρίτη, ίσως κάτι πολύ σύντομα που θέλω να σας πω, είναι το εξής. Μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, από το 2013 και μετά, θα ήθελα να τονίσω εγώ τα εξής τρία, που είναι και προτεραιότητες. Πρώτον, το δημογραφικό πρόβλημα βλέπουμε νέες δημογραφικές ανισορροπίες μέσα στην Ευρώπη και έχουμε και φαινόμενα άτακτης ε, μετανάστευσης και γύρανσης του πληθυσμού που από ε, περιφέρεια σε περιφέρεια της Ευρώπης διαφέρει η κατάσταση και θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Στη συνέχεια έχουμε το πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης που και αυτό είναι ένα στοιχείο κοινωνικής ταραχής και αταξίας. Και αυτό θα πρέπει να μας ε, οδηγήσει στην ανάγκη εξυγχρονισμού του ε, εργασιακού πλαισίου που διαθέτουμε. Και ένα τρίτο σημείο είναι το εξής. Για να υπάρχει κοινωνική συνοχή θα πρέπει να υπάρχει και συνοχή εδαφική. Δηλαδή η κινητικότητα στην Ευρώπη μέσω της βελτίωσης ε, των υποδομών, μεταφορών, των επικοινωνιών κτλ. θα πρέπει να είναι αποφασιστική σημασία. Και τέλος, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Κατά την άποψή μου, η επιτυχία αυτής της νέας στρατηγικής για την ε, κοινωνική συνοχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον καλύτερο και μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των εθνικών πολιτικών ε, κοινωνικής συνοχής και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχει λυθεί ακόμα, που εκκρεμεί. Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες. Και δεν μπορεί να είναι το Ταμείο Συνοχή ένα κουμπαρά και κάθε κράτο μέλο να αντλεί τα κονδύλια που χρειάζεται για να κάνει ό,τι του καπνίσει στη τελική ανάλυση. Και συγγνώμη που το λέω έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπροάζ Λεκ, ε, Ευρωβουλευτή από την Γαλλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση είναι πάρα πολύ επίκαιρη και σκόπιμη και δεν θέλω να επανέλθω στα σημεία που η Επιτροπή μας θεωρεί σημαντικά για την Ευρώπη, για την πολιτική συνοχής. Θα ήθελα ίσως να επιμείνω στο γεγονός ότι η κρίση που ζούμε σήμερα μας οδηγεί στο να ε, αμφισβητήσουμε και πάλι γενικώ ε, τις ε, κατευθύνες γραμμές και την πηξίδα που είχαμε μέχρι τώρα στην οικονομική και στη χρηματοπιστωτική κατάσταση γνωρίζουμε ποια είναι η κρίση βλέπουμε τώρα και τεράστια κοινωνική κρίση τα θέματα τα περιφερειακά και τα εδαφικά θα τα δούμε στο μέλλον με μεγάλη οξύτητα μπροστά μας ε, και όλα αυτά μας οδηγούν ε, στο να έχουμε μια νέα προσέγγιση και θεώρηση της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Θα ήθελα λίγο να επιμείνω σε αυτό λέγοντας ε, στη Σουηδή συνάδελφό μου επιτρέπει ότι θα χρειαστεί λίγο να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε και αυτά που λέμε. Ότι έχουμε ε, χαράξει ένα δρόμο που είναι κούρσα στην ανταγωνιστικότητα, ανοίγουμε τις αγορές, μειώνουμε τη φορολογία. Αυτό λίγο έχει αρχίσει να κλονίζεται. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε. Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν έχουμε διαπιστώσει ε, ότι Υπάρχει κάποια σύγκληση αρκετά πετυχημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το ταξί των κρατών μελών, παλιών ή νέων. Πείτε τα όπως θέλετε. Αλλά υπάρχουν ακόμα στρεβλώσεις και διαφορές σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο. Περισσότερο σε κάποιες χώρες από ό,τι σε κάποιες άλλες. Γι' αυτό είπαμε ότι χρειάζεται μια πραγματική πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι επανεθνικοποίηση αρκεί να δει κανείς ποια προβλήματα θέτουν ε, τα εθνικά σχέδια που είτε προετοιμάζονται είτε ε, υλοποιούνται για να απαντήσουμε σήμερα στην κρίση. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Ε, είναι προφανές αυτό. Και να επιμείνω σε κάτι που απασχολεί την Επιτροπή μας Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Γενικέ Διευθυντά, και κάτι το οποίο θα απασχολήσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Γι' αυτό είναι η, η Λισαβόνα. Δεν θέλω να γίνει σύγχυση ανάμεσα ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας που περιμένουμε διακαώς με τεράστια ανυπομονησία και τη στρατηγική της Λισαβόνας που είναι άλλο πράγμα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η στρατηγική της Λισαβόνας είναι μια στρατηγική που ακόμα δεν έχει ευθυγραμμιστεί με ε, την κοινωνική συνοχή και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και μπορεί ενδεχομένως να μας οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου οι Ευρωπαίοι να απομακρυνθούν ακόμα περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που καταρχάς δική τους ένωση είναι των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό το θέμα νομίζω θα τεθεί πάρα πολύ έντονα το 2013. Μερικοί από εμά ε, δεν θα είμαστε πια εδώ μεταξύ αυτών και εγώ. Ε, πάντως ε, δουλεύουμε προς την κατεύθυνση της πολιτικής συνοχής έτσι με μεγάλο πάθος γιατί είναι σημαντικό αυτό για το μέλλον για να ανταποκριθούμε και να απαντήσουμε στις σημερινές προκλήσεις, στις μελλοντικές προκλήσεις που είναι τεράστιες και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε απολύτως έτοιμοι, πανέτοιμοι για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε πει ότι είναι βασικό στόχος της Ένωσης η περιφερειακή συνοχή, θα πρέπει να έχουμε και τη λευκή βίβλο και να είμαστε ε, αμέσως επιχειρησιακοί, λειτουργικοί από την πρώτη μέρα. Και να είμαστε και έτοιμοι βεβαίως για να απαντήσουμε σε όλα αυτά και δημοσιονομικά και επί της ουσίας. Τελειώνω λέγοντας σύντομα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο σε ένα τόσο αποφασιστικό θέμα για το μέλλον που είναι η κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να το αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει αυτό και ε, στην ε, εδαφική συνοχή, στο μέλλον των περιφερειών μας. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, άλλες μεγάλες περιφερειακές ενώσεις ε, θα μας ξεπεράσουν στον πλανήτη. Και υπάρχει φοβαρός κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαλυθεί ή να αποδιοργανωθεί μεταξύ διαφόρων οργανισμών, φτωχοί, πλούσιοι, πόλεις, περιφέρειες, απομακρυσμένες κεντρικές περιοχές, ο καθένας να τραβάει προς την κατεύθυνσή του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Βουλής της Λιθουανίας, είναι ο κύριος Βιταούτας Κουρπουβέσας. Συγγνώμη αν δεν είπα σωστά το όνομά σας, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ καταρχήν για τη σύγκληση της παρούσας συνάντησης. Σας ευχαριστώ για την ανοιχτή αυτή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον της. στην ε, ε, ε, Λιθουανία συντονίζονται καλά μεταξύ τους η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, η εθνική και η τοπική πολιτική. Και σκοπό έχει τη γεφύρωση των χασμάτων μεταξύ των περιφερειών από οικονομικής και κοινωνικής πλευράς. για να ε, εφαρμοστεί σωστά η πολιτική αυτή από το 2007 μέχρι το 2013 ε, πρέπει να πληρούνται κάποιες ε, προϋποθέσεις. Έχουν αναπτυχθεί περιφερειακά συστήματα. Μπορεί όμως μετά το 2013 να πρέπει να αλλάξουμε τα, συστήματα λόγω, της, λόγω μιας πιθανής μεταρρύθμισης ότι, πιστεύουμε ότι οι πιο αδύναμες ε, περιφέρειες ε, θα πρέπει να ε, βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει το πιο σημαντικό κριτήριο να είναι το ΑΕΠ ανα, κατά κεφαλή για να καθορίσουμε ποιες ε, περιφέρειες ε, δεν είναι αρκετά αναπτυγμένες. Θα πρέπει η πολιτική αυτή να ενισχύσει την αλληλεγγύη ανάμεσα στο, στα κράτη-μέλη. Οι τρεις βασικοί στόχοι, η σύγκληση, η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση, θα πρέπει να παραμείνουν και στο μέλλον. Ε, Έχουμε νέες προκλήσεις, ε, τι ε, δημογραφικές αλλαγές, ε, την παγκοσμιοποίηση, την αλλαγή του κλίματος, την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Πρέπει να πραγματοποιηθεί συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα πρέπει όμως η νέα συζήτηση αυτή να επισκιάσει τους βασικούς ε, στόχους της πολιτικής συνοχής. Η Λιθουανία στηρίζει την, ε, το συσχετισμό τη ε, περιφερειακής της πολιτικής συνοχής και της πολιτική της Λισαβόνας. Επιμένουμε όμως η εφαρμογή των δύο αυτών προγραμμάτων να παραμένει διακριτή στα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε επενδύσεις ε, στην υγεία, την ε, ε, εκπαίδευση, την έρευνα και τις κοινωνικές δομές. Αυτά δεν ανήκουν στην πολιτική της Λισαβόνας. Στην πράσινη βίβλο του Θηνοπόρου του 2008 η Κομισιόν τονίζει τη σημασία των θεμάτων αυτών για τους πολίτες. Θα πρέπει να ε, ελεγχθούν οι διοικητικές ε, δομές ε, και οι μηχανισμοί ελέγχου. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στις μελέτες αντικτύπου. Η διαρθρωτική βοήθεια θα πρέπει να προσανατολίζεται στα αποτελέσματα. Ήδη εξετάζουμε τις, ε, τους μακροπρόθεσμους ε, στόχους μας ε, και τα μέσα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να τους πετύχουμε. Η πολιτική συνοχής, λόγω της σημασίας της και των στόχων που ήδη έχουν επιτευχθεί, θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί σημαντική πολιτική της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Yes, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πιμέντα από την Πορτογαλία. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την πεποίθησή μου ότι οι πολιτικές συνοχής της Ένωσης είναι ένας βασικός πυλώνας της ίδιας της διαδικασία ολοκλήρωσης και γι' αυτό και αποκτούν έναν θεμελιώδη ρόλο στην μείωση των ε, διαφορών μεταξύ των περιφερειών και γι' αυτό και θα πρέπει και να συνεχιστούν μετά από το 2013 και γι' αυτό το λόγο και βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Γνωρίζουμε πως υπάρχει μια προφανή σε σχέση μεταξύ των ευρωσκεπτικιστών και της αύξησης ε, των διαφορών μεταξύ των περιφερειών και γι' αυτό και δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε τις πολιτικές ε, περιφερειακής ανάπτυξης για να στηρίξουμε την ίδια την νομιμότητα αυτών. Είμαστε επεπισμένοι ότι η πρόκληση θα είναι να συνεχίσουμε να προωθούμε την σύγκληση ανάμεσα στις ε, περιφέρειες, περιορίζοντας ε, τις διαφορές ανάπτυξης. Γνωρίζουμε πως σήμερα υπάρχουν περιφέρειες που πέρασαν από το στόχο 1 στον στόχο 2, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης και οι ίδιες βλέπουν την ανάπτυξή τους και την, το πιμπ τους, να, το ΑΕΠ να μειώνεται. Δηλαδή, είτε βρίσκονται στο στόχο 1, είτε βρίσκονται στο στόχο 2, υπάρχουν κοινέ προκλήσεις ε, στο σημερινό κόσμο. Γι' αυτό και θα υπάρχουν περιφέρειες όπου χρειάζεται περισσότερο να γίνουν επενδύσει στι υποδομέ από ό,τι σε άλλε, αλλά υπάρχουν και άλλε ε, περιφέρειες που θα χρειαστεί να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικέ και άρα να επενδύσουν στην οικονομία τη γνώση, στην καινοτομία και ούτω καθεξής. Δηλαδή, βασικά θα ε, πρόκειται για ένα συμπλήρωμα της της Λισαβόνας και γνωρίζουμε πως όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με βάση την βιωσιμότητα του κάθε προγράμματος, δηλαδή αυτό σημαίνει πως πρόκειται για μια οικονομία που θα βασίζεται στο σεβασμό του πλανήτη. Και είναι πεποίθησή μας πως οι προκλήσεις αυτές θα περάσουν από μια σύνδεση μεταξύ των πολιτικών ε, ε, συνοχής και των εθνικών πολιτικών. Ε, δηλαδή θα πρέπει εδώ να πούμε ότι θα πρέπει να γίνει συνδυασμός προσπαθειών ανάμεσα στα κεφάλαια τα, της συνοχής και άλλα μέσα ώστε όλα μαζί σε συνδυασμό να προωθήσουν προς την ανάπτυξη, την αρμονική των περιφερειών. Εγώ είμαι πεπισμένη και ήδη αναφέρθηκε αυτό από ορισμένους ότι το, οι της αναδιάρθρωσης θα πρέπει να απογραφειοκρατικοποιηθεί γιατί γνωρίζουμε πως ε, ταυτίζεται ανέκαθεν ε, με τις ε, κοινοτικές γραφειοκρατικές δομές ενώ εμείς χρειάζεται να είμαστε ταχείς και καινοτόμοι ταυτόχρονα. Και έχω την εμπειρία ότι το πακέτο αυτό, το οποίο ε, στόχο έχει να απλοποιήσει τους κανόνες εφαρμογής ε, των πολιτικών συνοχής, θα πρέπει να έχει ταυτόχρονα και στόχο την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών συνοχής. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα γρήγορα αλλά και σωστά. Γι' αυτό και ελπίζω ότι η ανάλυση της απλοποίησης θα είναι σημαντική βέβαια, αλλά ε, θα είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε ότι και η διαφάνεια είναι εξίσου σημαντική και πρέπει να μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε την λιγότερη γραφειοκρατία με την μεγαλύτερη διαφάνεια. Εάν δεν υπάρχει σωστή πολιτική συνοχή, δεν θα υπάρχει και ένωση. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κύριο Βανίστελ Ρόι, που είναι ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μάλιστα. Πολύ καλό είναι που παίρνουμε τώρα λίγο χρόνο και αφιερώνουμε ε, ε, στη συζήτηση παραμονές της καινούργιας θητείας για να δούμε πού βρισκόμαστε. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συζητάμε πολύ, αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θυμάμαι όταν συζητούσαμε το οικονομικό πλαίσιο και γίνεται κυρίως λόγος πάντα για τα λεφτά και ποτέ για το περιεχόμενο. Και επειδή είναι πάντα οι επταετής οι προγραμματικές περίοδοι, είναι αρκετό διάστημα για να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις για το μέλλον και από τη σκοπιά αυτή να τα βλέπουμε τα πράγματα, όχι από το τι έγινε στο παρελθόν. Και εγώ πιστεύω, ακράδαντο, ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί η πολιτική. Και Είπε ο πρόεδρος ας ξεκινήσουμε από την αφετηρία ότι δεν είναι απολύτως απαραίτητο και δεδομένο ότι θα διατηρηθεί ο στόχος 2. Καλό είναι αυτό να το συζητάμε. Δεν μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε μεγάλους προϋπολογισμούς που διπλασιάζονται πολλές φορές και όλο περισσότερο δίνονται σε έρευνα και ανάπτυξη ας πούμε, χωρίς ταυτόχρονα να έχουμε την οποιαδήποτε σύνδεση ε, με την περιφερειακή πολιτική. Μιλάμε για ανταγωνιστικότητα ε, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, από τις περιφέρειες, από τη συνοχή. Ενισχύθηκαν τα τελευταία 20-25 χρόνια οι περιφέρειες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια νέα σχέση ανάμεσα στα χρήματα αυτά που δίνονται ε, υπέρ της αριστείας από τις Βρυξέλλες και περιμένω από τα 54 δις την επόμενη φορά να είναι 100 δις, εντάξει δεν πειράζει, αλλά αυτά θα πρέπει να καταλήγουν στις περιφέρειες, στα λεγόμενα clusters, σε διάφορους πόλους. Ε, αυτό το λέει και η πράσινη βίβλος. Ε, Βεβαίω από τη μια λέω ναι κατά της συγκέντρωσης, γιατί δεν θέλω να υπάρχει συγκέντρωση, αλλά αν δεν δώσουμε απάντηση στο πώς μεταφέρουμε τη γνώση μεταξύ των περιφερειών ε, στην Ευρώπη δεν θα έχουμε την απάντηση που χρειαζόμαστε. Είναι νέοι καιροί, χρειάζονται νέες απαντήσεις. Ε, βλέπουμε και την κρίση που ζούμε τελευταία, την οικονομική. Σωστά μας είπε εκπρόσωπος της Σουηδίας ότι θέλουμε νέες απαντήσεις στα νέα προβλήματα. Γι' αυτό πιστεύω καλό θα ήταν εσείς τώρα να κάνετε τη συζήτηση στα εθνικά κοινοβούλια και μην περιμένετε την πέμπτη έκθεση συνοχής και την πρόταση για το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Διότι αυτή είναι η τελική συζήτηση, αλλά δεν θα έχουμε κάνει την προκαταρκτική χωρίς να υπάρχει ένα καλό υποκείμενο όραμα για το πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον. Και καλά κάνουμε και το συζητάμε σήμερα λοιπόν εδώ. Ε, αν μου επιτρέπετε ένα σημαντικό ακόμα στο Κοινοβούλιο εδώ έχουμε βέβαια πολιτικές ομάδες. Εγώ είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Την περασμένη χρονιά σκεφτήκαμε πάρα πολύ αυτά τα θέματα, μας προβλημάτισαν και φτιάξαμε ένα φυλάδιο και είναι σημαντική η πολιτική συνοχή. Θα πρέπει να συνεχιστεί η σύγκληση και το τονίζω, εντάξει, αλλά θα πρέπει για το στόχο 2 να έχουμε νέες ε, προτάσεις θα πρέπει να, με δημιουργικότητα να το συζητήσουμε και να αξιοποιήσουμε και τις δικές σας συζητήσεις στα Εθνικά Κοινοβούλια. Και τέλος, για το στόχο 3, τη διασυνοριακή διαπεριφερειακή συνεργασία, θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή εκεί. Είναι υπερβολικά περιθωριοποιημένο αυτό στον προϋπολογισμό. Και τελικά δεν πάει καλά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται αυτό όχι μόνο στα εξωτερικά σύνορα αλλά και στις νέες περιφέρειες, ακούσαμε για τις χώρες της Βαλτικής, έτσι ώστε κάποια κράτη-μέλη που είναι πολύ μικρά να μπορούν να υποφιλούνται ας πούμε ε, και από την αριστεία, την τεχνολογική και από την οικολογική ποιότητα ας πούμε ο Δούναβης και κάποιες άλλες ε, περιφέρειες που υπάρχει συνεργασία θα πρέπει αυτό να γίνεται διασυνοριακά εντός της Ένωσης, όχι μόνο στα εξωτερικά σύνορα. Και εδώ χρειάζεται ε, ε, νέα προσέγγιση. Σας συνιστώ αυτό το φυλάδιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Διατίθεται σε τέσσερις γλώσσες. Πάρτε το μαζί σας, το διαβάστε. Είναι πολύ χρήσιμο για τη συζήτηση. Thank you very much. like to give Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Θαλασσινός, Θαλασσινός από το, την Ελληνική Βουλή. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ε, Πρόεδρε, Πράγματι θα, θα επισημάνω και εγώ την σπουδαιότητα της σημερινής κοινή συνεδρίασης γιατί το θέμα της πολιτικής της συνοχής είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και απασχολεί όλους μας σε επίπεδο ε, εθνικό, περιφερειακό και υπερεθνικό. Η πολιτική της συνοχής στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει πλέον σαφές περιεχόμενο και αποτελεί ένα βασικό και αυτόνομο πολιτικό πυλώνα που λειτουργεί οριζόντια και υποστηρικτικά προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πολιτικές. Πιστεύω ότι κομβικό σημείο σε αυτή την πολιτική πρέπει να είναι η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων, ανισότητες που είναι πολύ πιθανό να ενταθούν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης όσο και της πιθανής στρέβλωσης του διεθνούς ανταγωνισμού. Εκτιμώ κύριε Πρόεδρε ότι, και κύριοι συνάδελφοι ότι ειδικά για τις νησιωτικές, ορεινές και γενικά απομονωμένες περιοχές της Ευρώπης πρέπει να ληφθεί μέρημνα για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανισότητες και να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν και τις οποίες, οι οποίες επισημάνθηκαν. Το λέω αυτό και με πλήρη γνώση αν θέλετε διότι κατάγομαι και εκλέγομαι σε μια νησιωτική περιοχή της Ελλάδας η οποία είναι ταυτόχρονα και ορεινή και αρκετά απομακρυσμένη από το κέντρο. Για μας στην Ελλάδα φαντάζομαι και για τις άλλες χώρες είναι σημαντική εξέλιξη ενσωμάτωση της χωρικής συνιστώσας στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής γεγονός που μπορεί να οδηγήσει για παράδειγμα σε μια ενιαία πολιτική για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να ενδυναμωθεί κυρίως προς τις εξής κατευθύνσεις. Χρειάζεται να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης των ενδοπεριφερειακών οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων να υπάρξει συντονισμός ως προς τις τομεακές πολιτικές σε έρευνα, καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, περιβάλλον, περαιτέρω εξειδίκευση στα θέματα της χωρικής διάστασης και αντιμετώπιση των κοινών μειονεκτημάτων των απομακρυσμένων περιοχών, νησιά, ορεινές περιοχές, αρεοκατοικημένες περιοχές, να δούμε το ζήτημα της παράνομης εισρωής μεταναστών που πλήττει τα θαλάσσια σύνορά μας, να βρεθούν τρόποι μέτρησης των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ώστε να κρίνουμε και τα αποτελέσματα των εφαρμοσμένων πολιτικών. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών και πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατό περιθώριο για την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών. Σας ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Πολωνική Βουλή. Ο κ. Ιωσόφ Όρτελ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα θερμά να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα να συμμετέχω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο ρόλος της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εξαιρετικά σημαντικός. Στη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε, τη, να μάλλον να έχουμε υπόψη μας την ε, σύγχρονη οικονομική κατάσταση και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις ε, για την περίοδο μετά το 2013. Για παράδειγμα, Νομίζω ότι μπορεί να καταλήξουμε σε δυσκολίες στην ασφάλεια ανεφοδιασμού ενέργεια μετά από την ε, οικονομική αυτή κρίση βέβαια μπορεί να έχουμε και ένα ακόμα μεγαλύτερο κενό, μάλλον διαφορά αναπτυξιακή ανάμεσά μας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε για το μέλλον. Φυσικά η οικονομική κρίση είναι ένα πρόβλημα, ωστόσο ε, στο φως της ε, πολιτικής συνοχής αποτελεί μια πρόκληση, μια ευκαιρία ώστε να μπορέσουμε να ε, δώσουμε νέους προσανατολισμούς σε αυτή την πολιτική. Η συζήτηση που γίνεται στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στις διάφορες συναντήσεις, διάφορα σώματα δείχνει ότι θα πρέπει όντως να συνεχίσουμε με την πολιτική συνοχή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ε, διαδικασίας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ωστόσο οι αρχές και οι στόχοι απαιτούν διόρθωση όπως επίσης απαιτεί διόρθωση του σύστημα εφαρμογής. Οι πολιτικοί στόχοι, οι προτεραιότητες θα πρέπει να προσδιοριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε η πολιτική να εστιάζει την προσοχή σε ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό στόχων και προτεραιοτήτων. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη ανάπτυξη στην κοινότητα, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης και θα πρέπει να προσπαθήσει να περιορίσει τις ανισότητες ανάμεσα στους ε, φτωχού, στις φτωχότερες και τις πλουσιότερες περιοχές. Θα πρέπει να αποτελεί ένα μέσο αλληλεγγύης ε, Καλό θα ήταν να εξετάσουμε και το ειδικό λειτουργικό πρόγραμμα για τις πέντε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Πολωνίας, καθώς και άλλα ειδικευμένα προγράμματα αυτού του τύπου. Και φυσικά, πολιτική συνοχής θα πρέπει να εξεταστεί ως μια οριζόντια πολιτική υπέρ της ανάπτυξης. Δεδομένου ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να συνδυάζει τις διάφορες ε, συνιστώσεις ε, της προσπάθειας υπέρ της ανάπτυξης θα πρέπει να σκεφτούμε και την κατάργηση των φραγμών ανάμεσα στα διάφορα ταμεία. Ίσως ε, να πρέπει να ενσωματωθεί η στήριξη της ανάπτυξης πέθρου στην πολιτική συνοχή. Πιστεύω πως όλοι γνωρίζουμε πώς γίνεται ο προγραμματισμός στην πράξη, πώς οι διαχωριστικές γραμμές καθορίζονται. και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πάντοτε απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στις πράξεις και στους ε, στόχους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων σε προβλήματα, αλλά και σε προβλήματα κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ελέγχου. Εγώ πιστεύω πως ολόκληρη η πολιτική θα μπορούσε να ακολουθήσει μια πιο αποτελεσματική κατεύθυνση. Σαφώς και καλωσορίζω το γεγονός ότι... Ε, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για το χρήμα που δίνουμε σε αυτή την πολιτική. Μιλάμε περισσότερο και είναι πιο σημαντικό αυτό να μιλήσουμε για τις αρχές και για τις κατευθύνσεις. Ωστόσο, στο μέλλον δεν πρέπει να υπάρξει και μείωση των πόρων που απευθύνονται στη πολιτική συνοχή. Οι τρεις διαστάσεις θα πρέπει να διατηρηθούν. Θα, πρέπει μια πολιτική, η πολιτική αυτή που θα ε, σχεδιάσουμε να επιτύχει και αυτό σημαίνει επαρκείς αξιόπιστους δείκτες ανάπτυξης. Δεν πρέπει να περιοριστούμε στις οικονομικές παραμέτρους. Θα πρέπει να έχουμε δημογραφικές παραμέτρους, να σκεφτούμε την ε, κοινωνική, την, ε, και τις χωρικές παραμέτρους επίσης. Σας ευχαριστώ γερουσιαστά Όρτελ και τώρα καλό τον κύριο Γιανόφσκι που είναι ε, ευρωβουλευτής από την Πολωνία να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. ενδιαφέρουσα από συζήτηση. Πόσες φορές σήμερα το απόγευμα ακούσαμε τη λέξη κρίση. Δεν είναι όμως ε, καιρός για πανικό ή για χάος. Είναι η κατάλληλη στιγμή για ψύχρεμη, ήρεμη ε, ήρεμο προβληματισμό. Να σας θυμίσω τον πιλότο που ασφαλώς προσγείωσε ένα αεροσκάφος στον ποταμό Χάτσον σώζοντας όλους τους επιβάτες και το αεροσκάφος. Αυτή του είδους την ψυχραιμία χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ε, παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή ναι. σε όλα αυτά ακούγονται πολύ καλά, αλλά μην ξεχνάμε το πόσιμο νερό για το μέλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμπεριλάβατε στον προβληματισμό σας. Σε σχέση τώρα με το μέλλον της πολιτικής συνοχής, θα πρέπει να σκεφτούμε τα αποτελέσματα της σύγχρονης πολιτικής συνοχής. Δεν ξέρω αν αυτό προλαβαίνουμε να το κάνουμε πριν από τις ευρωεκλογέ, αλλά θα ήταν καλό για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθήσουν ή να, στείλουν, να πάρουν πληροφορίες, σε πάση περιπτώσει, μια επιστολή που σαφώ θα τους εξηγεί πώ δαπανήθηκαν τα χρήματα. Νομίζω πως τα χρήματα έχουν δαπανηθεί πολύ καλά. Μια, ένα σχετικά μικρό ποσό έχει οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι ένα ευρώ στο πλαίσιο μια σωστά προγραμματισμένης πολιτικής. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει εξάλλου αντίφαση ανάμεσα στις υποδομές και στην κοινοτομία. Και νομίζω πως θα ήταν ε, λάθος το να κάνουμε ε, το να τα διαχωρίσουμε στο περιβάλλον. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να, κάνουν στην ενέργεια, να γίνουν στην ενέργεια επίσης, αλλά πάνω απ' όλα η συνοχή θα πρέπει να, λαμβάνει, να είναι προ όφελος όλων των 500 εκατομμυρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στην παιδεία, στην ποιότητα ζωής, στην υγειονομική περίθαλψη και ούτω καθεξής. Εάν δείτε πώς έχει τώρα η κατάσταση, υπάρχει δεκαπλάσια διαφορά στο κατακεφαλήνα έπος ανάμεσα στην πλουσιότερη και στη φτωχότερη περιφέρεια και είναι τεράστια η διαφορά αυτή. Γι' αυτό και θα πρέπει να στηρίξουμε τους καινοτόμους, τους, τοπικού, τους τοπικούς, ε, τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο σε έναν εκπρόσωπο του Ισπανικού Κοινοβούλιο. Την κυρία Μέριτσελ Μπάτετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, ε, όνομα είναι και αυτό που έχω. Είναι περίπλοκο και στην ίδια μου τη χώρα κάνουν λάθος. Οπότε δεν φταίτε εσείς. Έχω εγώ. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία και θα ήθελα να εθαρρύνω την Τσεχική Προεδρία να κάνει διάφορα σεμινάρια σε διάφορα επίπεδα και εδώ και αλλού. Θα ήθελα εγώ να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Άνερ, ο Γενικός Διευθυντής, όταν μας είπε ότι όλα τα προβλήματα του μέλλοντος, που είναι βεβαίως ε, παγκόσμια, κοινωνικός αποκλεισμός, δημογραφικές αλλαγές, ε, μεταναστευτικά ρεύματα, θέματα ενέργειας, θέματα νερού επίσης. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουν επιπτώσεις λέει στην πολιτική συνοχής. Εντάξει. Θα πρέπει να έχουμε όμως στο μυαλό μας ότι και η πολιτική συνοχής θα έχει επιπτώσεις σε αυτές τις προκλήσεις του μέλλοντος, διότι σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από το πώς ορίζουμε αυτές τις δημόσιες πολιτικές. Όχι μόνο συνοχής, όλες τις πολιτικές, επαναλαμβάνω, όλες τις πολιτικές. Ποιε θα είναι οι προτεραιότητες ε, και πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα ή λιγότερο καλά αυτές τις προκλήσεις. σε κάθε περίπτωση αυτές οι προκλήσεις έχουν μια διάσταση υπερεθνική, υπερκρατική, ξεπερνάει τα κρατημέλη. Και ξεπερνάει και την Ευρώπη την ίδια. Ε, επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί σε εθνικό πλαίσιο. Τις λύσεις λοιπόν δεν μπορούμε να τις δώσουμε τοπικά ο καθένας ξεχωριστά. Θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι οι πολιτικές μας για να διαχειριστούμε αυτή την πολυπλοκότητα. Ε, σε κάθε περίπτωση ε, θα πρέπει αυτό να έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων Ευρώπη, κράτη, περιφέρειες και οτά ακόμα οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και επίσης θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία, συντονισμός μεταξύ των διαφόρων πολιτικών οι πολιτικές δηλαδή, ενώ όχι τους πολιτικούς, που θα πρέπει και σε κοινοτικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο να είναι συντονισμένες. Λοιπόν, ειλικρινά γι' αυτό ε, όλες οι προτάσεις περί επανεθνικοποίησης και τα λοιπά, και θέλω να μιλήσω και για τον Ιταλό συνάδελφο που αναφέρθηκε σε αυτό, άμεσα και αντιτάχθηκε σε αυτή την επανεθνικοποίηση, θέλω και εγώ να πω πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή, ότι θα ήταν οπισθοδρόμηση η επανεθνικοποίηση. Οι πολιτικές της συνοχής δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι επανεθνικοποιημένες, δεν μας οδηγούν καθόλου ούτε στη συλλογική ε, επιτυχία, αλλά ούτε στη μεμονωμένη επιτυχία κανενός. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο πειρασμός, ο καθένας να προστατεύει το δικό του τη γειτονιά του, το χωριό του να περιχαρακωθεί σε ένα κλειστό κύτταρο ομοιογενές από τον έξω κόσμο. Αυτό δεν λύνει τίποτα, ε, ειδικά στη σημερινή εποχή της κρίσης. Αλλά και την κρίση να μην είχαμε δεν θα ήταν θετικό κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο θετικό δεν θα ήταν, αλλά αντιτίθεται και στις αρχές μας τις ίδιες επιτίθεται στην ίδια την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρχές μας, με βάση τις οποίες όλα αυτά τα χρόνια οικοδομούμε τούτη εδώ την Ένωση. Είναι σημαντικό και τελειώνω με αυτό, η Ένωση να θεωρεί τον εαυτό της παγκόσμιο πρωταγωνιστή και να δράω ως τέτοια και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εργαζόμαστε όλοι μαζί από κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, now I would like to give the floor the uh, representative of Romanian Senate. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Γερουσίας της Ρουμανίας, τον κύριο Φίλιπ Πέτρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εδώ είμαι. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέρφους από την Επιτροπή Ρέτζι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα καθότι όπως ξέρετε μέχρι πριν δύο μήνες ήμουν μέλος της Επιτροπής αυτής. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής ήταν ένα από τα βασικά θέματα της Επιτροπής Ρέτζι, Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής είναι ένα μέσο που βοηθάει την Ένωση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια συζήτηση, μια τέτοια συνάντηση όπως αυτή που έχουμε σήμερα, πιστεύω ότι θα πρέπει να επαναληφθεί στο μέλλον. Ενδεχομένως με περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε τα προβλήματα αυτά, ιδιαίτερα καθότι τα επόμενα χρόνια, οι επόμενοι μήνες, τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι εύκολα. Και ακριβώς επειδή τα εθνικά κοινοβούλια έχουν και λόγο όσον αφορά τη μεταφορά των ευρωπαϊκών προτύπων σε εθνικό δίκαιο. Να σας θυμίσω τις συζητήσεις που είχαμε στην Επιτροπή Ρέτζι πέρσι σχετικά με τον ορισμό της συνοχής. Στο παρόν πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, όπως είπε ο συνάδελφος Γιακουμπόσκι, η κρίση βρίσκεται εδώ, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε. Στο πλαίσιο αυτό να κάνω κάποιες προτάσεις εκ μέρους της ε, Ρουμάνικης Γερουσίας. Τρεις προτάσεις έχουμε ουσιαστικά. Διατήρηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, να το διατηρήσουμε ως βασικό ε, μέσο δράσης όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής για να πετύχουμε πολιτική αποτελεσματικότητα μέσω της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας των δράσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε κυρίως τη μετακίνηση του ε, ταμείου αυτού ε, ώστε να μην ε, υπόκειται πια στα διαφορετικά ταμεία. Επίσης θα πρέπει να βρούμε έναν κοινό μηχανισμό συνεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήταν επίσης σημαντικό να συγκεντρώσουμε τους οικονομικούς πόρους της πολιτικής συνοχής σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων. Σκέφτομαι ενδεχομένως μια θεματική συγκέντρωση, κάποιους ε, τομείς ανάπτυξης, κάτι που θα βοηθούσε και την αύξηση της απασχόλησης. Για τη Ρουμανία, σημαντικό και δύσκολο θέμα, είναι το γεγονός ότι είμαστε ε, ε, χώρα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένων των ε, παγκοσμίων εξελίξεων η Ρουμανία θα βρεθεί σε δύσκολη θέση όσον αφορά τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ανατολικούς μας γειτόνους. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό να αναφέρω την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών εφαρμογής της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή της αναλογικότητας, να απλοποιήσουμε διαδικασίες ε, διαχείρισης και ελέγχου, ε, να απλοποιήσουμε τους κανόνες που έχουν να κάνουν με την κρατική ενίσχυση, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς όπως είναι ε, το περιβάλλον, η επαγγελματική κατάρτιση κλπ. Επίσης, η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τα διαρθρωτικά ταμεία. Ξέρω ότι αυτά ήταν θέματα που έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή Ρέτζη. Να προτείνω για άλλη μία φορά η πρωτοβουλία αυτή της Επιτροπής ε, Ρέτζη, αυτή η ανταλλαγή με τα Εθνικά Κοινοβούλια να συνεχιστεί. Ακόμα κι αν δεν απομένει πολύς χρόνος λόγω των επικείμενων ευρωεκλογών. Μετά από αυτό όμως ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για μελλοντικές συναντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, πολύ σωστά. Είσαστε εκπρόσωπος της ε, Γερουσίας, ε, δεν το είπα σωστά πριν. Ε, θα παρακαλούσα τώρα τον κύριο Γιώζεφ Βέρες από την Ουγγαρία να πάρει το λόγο από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με εκπλήσει κάπως. Αισθάνομαι λίγο σαν να κάνουμε, σαν να μην τρέχει τίποτα. Διανύουμε μια κρίση παγκόσμιας κλίμακας συζητάμε σε άλλες επιτροπές πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα κονδύλια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κράτη να ξεπεράσουν και να επιβιώσουν. Είμαστε βέβαιοι ότι το 2013 οι συνθήκες θα είναι οι ίδιες με τις σημερινές. Δεν νομίζω εγώ. Νομίζω πως πραγματικά πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας, την οποία περιμένουμε πώς και πώς, μπορεί ήδη να είναι πεπαλαιωμένη, ξεπερασμένη όταν θα αρχίσει να ισχύει. Χρειαζόμαστε ένα άλλου είδους ευρωπαϊκή συνεργασία για να ξεπεράσουμε την κρίση στην οποία έχουμε βουτυχτεί όλοι. Χρειαζόμαστε μια πολύ πιο αποτελεσματική περιφερειακή πολιτική και λείπει η δημιουργικότητα. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε τη δυνατότητα στις περιφέρειες να ξεπεράσουν την κρίση. Η πολιτική συνοχή σε αυτό που τώρα συζητάμε έχω πολύ σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να απαντήσει όλα αυτά τα ερωτήματα. Το βασικό ζήτημα είναι αν πραγματικά πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων αυτό που βάζουμε δηλαδή ως βασικό πολιτικό στόχο ισχύει. Τουλάχιστον από το 1995 γνωρίζουμε ότι ε, παγκοσμίω γύρω στο 20% του εργατικού δυναμικού παγκοσμίου θα μπορεί να πληρεί τις ανάγκες της ανθρωπότητας. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει στο μέλλον να βάζουμε στόχο να βρούμε δουλειά στο 80% του απασχολητέου εργατικού δυναμικού. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη με αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και φοβάμαι πως η κρίση την οποία διανύουμε τώρα και που φαίνεται να προσθέτει, να τελειώνει μάλλον 300 χρόνια της βιομηχανικής κοινωνίας, ε, δεν έχουμε Ωστόσο, απαντήσεις, ποια είναι η κοινωνία στην οποία προχωράμε, η κοινωνία της γνώσης και ποιο είναι η μεταβατική περίοδος αυτή τη στιγμή. Πώς λοιπόν, εφόσον δεν ξέρουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του να διατηρήσουμε το εργατικό μας δυναμικό μαζί με βιώσιμες και ε, δυνατότητες απασχόλησης. Μιλάμε για αλληλεγγύη και ε, δυναμικό. Το βασικό ζήτημα είναι αν τα ταμεία συνοχής δίνουν δυναμισμό μόνο για τους δικαιούχους ή αν δίνουν τουλάχιστον τον ίδιο δυναμισμό και στις χώρες. Στόχος αυτό είναι και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν συζητάμε ως ήθιστε για το ποιος θα πληρώσει τα πιο πολλά και ποιος θα πληρώσει τα λιγότερα. Κάτι ακόμα και ίσως να μην είναι και πολύ ευγενικό να το θίξουμε, αλλά είναι ένα πραγματικό πολιτικό ζήτημα και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Πραγματικά πιστεύουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβιώσει με έναν προϋπολογισμό που είναι γύρω στο 1% του ΑΕΠ των εθνικών κρατών μελών, όταν όλοι οι ανταγωνιστές μας έχουν ε, ε, ε, τρεις-τέσσερις φορές μεγαλύτερο ε, μεγαλύτερης δυνατότητας. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει αυτή η ερώτηση, αλλά πρέπει να τη θέσουμε. Εγώ θαύμασα την εισήγηση του κύριου Διευθυντή, αλλά υπάρχουν δύο πράγματα στα οποία σίγουρα θα πω όχι. Δεν νομίζω πως τα κράτη, έθνη θα πρέπει, τα κράτη θα πρέπει να παίρνουν πιστώσεις για να χρηματοδοτήσουν τις περιφερειακές τους πολιτικές. Ε, ε, συγγνώμη, ότι θα πρέπει να επενεθούν τα κράτη-μέλη για την περιφερειακή τους πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενεθεί, γιατί εκείνη μπόρεσε να φτιάξει περιφερειακή πολιτική και να βρει τα κονδύλια που να έχει νόημα και να σημάνει τη διαφορά. Αν θέλουμε να παναπατρίσουμε την <laughs> περιφερειακή πολιτική, θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα, ποια θα είναι η διαφορά. Θα παίρνουν όλα στις δάφνες όπως προσπαθούν και τώρα να το κάνουν. Αυτό σε σχέση με την επανεθνικοποίηση της ε, περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Το πραγματικό θέμα είναι ότι αυτή η πολιτική συνοχή θα πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη και, να... και στοχοθετημένη ταυτόχρονα. Αλλά έχω σοβαρές αμφιβολίες για το αν ε, θα έχει κανένα πλεονέκτημα η πανεθνικοποίηση αυτής της πολιτικής. Αναφέρεται τώρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ναι, Πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τα επόμενα χρόνια. Είναι μεγάλο θέμα το πόσες θα επιβιώσουν ε, την κρίση που διανύουμε. Και ήδη είμαστε υποχρεωμένοι να επαναπροσδιορίσουμε το μερίδιο των χρημάτων που πρέπει να τους ε, δώσουμε άμεσα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ταυτόχρονα ε, φροντίζουμε το τραπεζικό σύστημα και τις πολυεθνικές, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει άμα δεν έχουμε δουλέψει αποτελεσματικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ξέρουμε πως χρειάζονται πάρα πολύ σε αυτού του είδους τη στήριξη και δεν είναι μόνο για τη δική τους επιβίωση. Το σημαντικό θέμα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σχετίζεται με το κατά πόσο ο τομέας των μικρομεσαίων εν γέννη μπορεί να είναι ανταγωνιστικό στο μέλλον και η στήριξη της επιχειρηματικότητας θα είναι ένας χρήσιμος παράγοντας και θα ήθελα να θίξω το θέμα της μεταφοράς γνώσης όσον αφορά την ε, ε, και την βελτιωμένη χρηματοδότηση. Αυτό που αναφέρεται για, το πράσινο, για την κίτρινη κάρτα για τα εθνικά κοινοβούλια είναι σημαντικό θέμα. Αλλά αν συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις πολιτικά μέσα στα παλιά πλαίσια, αυτό δεν βοηθά. Συγγνώμη που είμαι λίγο έτσι κάθετος, αλλά νομίζω πως εάν δεν βγούμε από τις παλιές μας ε, θέσεις, δεν έχουμε καμιά πιθανότητα, ούτε καν μετά από το 2013, να συνεχίσουμε. Ακόμα και αν πούμε ότι τα καταφέρουμε πάμε μέχρι το 2013. Θα θα ζητήσω μετά να μας απαντήσετε, κύριε Άνερα, αλλά όχι ακόμα. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βλάσακ, τον ε, Τσέχο Ευρωβουλευτή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Άκουσα προσεκτικά την ε, συζήτηση, όπως έχω ακούσει και προηγούμενες συζητήσεις ε, και μου είναι σαφές ότι κάθε ε, περιφέρεια έχει προβλήματα κάποιου τύπου. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται να γίνει η αναθεώρηση και ανάλυση της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να δούμε που λειτουργεί και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι η πολιτική συνοχή διατηρεί τη θέση της ε, στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό υπό το φως των μελλοντικών ε, αναγκών. Το 1 τρίτο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, πηγαίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Χρειαζόμαστε την ανταλλαγή απόψεων με εθνικά κοινοβούλια αλλά και με περιφερειακά και φυσικά και με τοπικές αρχές. Ε, πόλεις και χωριά. Και χάρηκα που άκουσα τον κύριο Άνερ και άλλους ε, και τον Επίτροπο στην Πράγα την Παρασκευή να μιλάει για συνεργασία και εταιρική σχέση. Χαίρομαι επίσης που κατά τη διάρκεια της εχικής Προεδρίας έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εκδηλώσεις ε, που ε, ασχολούνται ιδιαίτερα με το θέμα των αστικών περιοχών στη νέα εποχή. είναι οι λεγόμενες αστικές μέρες της Ευρώπης ε, την προηγούμενη Παρασκευή και Σάββατο και ε, πραγματοποιήθηκε και η πρώτη διάσκεψη των περιφερειών που λεγόταν ε, Czech Reg Days και ήταν η πρώτη φορά που οι περιφέρειες κατάφεραν να συνδυθούν μεταξύ τους. Υπό το, την ηγεσία της Νότιας Βοημίας συζήτησαν το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής. Το κύριο μήνυμα από όλες τις συζητήσεις αυτές ε, είναι η συνένεση σχετικά με το, την ανάγκη να καταλάβουμε ένα τον άλλον, να μιλάμε με τους ίδιους όρους. Πρέπει να, να συμφωνήσουμε τι ε, εννοούμε όταν μιλάμε για, για περιφερειακή πολιτική, τι εννοούμε όταν λέμε εδαφική πολιτική, τι λέμε όταν μιλάμε για αστική διάσταση. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας. Άλλο θέμα είναι το ότι θεσπίζουμε τα κριτήρια για τη χρήση των διαφθορτικών ταμείων σε διάφορα επίπεδα. Ξέρουμε όμως από πείρα ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει μια σειρά προϋποθέσεις, αυτές πολλαπλασιάζονται, διότι έχουμε μετά επιπλέον εθνικά κριτήρια και προϋποθέσεις και αυτά αναπτύσσονται και περαιτέρω σε τοπικό επίπεδο. Πιστεύω ότι η επικουρικότητα θα πρέπει να είναι η βασική αρχή, η πρωτεύουσα αρχή και ε, οι περιφέρειες θα πρέπει να υπαγορεύουν τους όρους. Ε, οι μεγάλες αστικές περιοχές που είναι υπεύθυνε για την εδαφική ε, διαχείριση και τον προγραμματισμό είναι σε θέση να στοχεύσουν τις δράσεις σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει στα πλαίσια της ε, παρούσας οικονομικής κρίσης είναι το όλο θέμα της πολιτικής ενισχύσεων. Ξέρουμε ότι η πολιτική συνοχής ε, χρηματοδοτείται με ενισχύσεις. Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη της Επιτροπής μας χρειάζεται να εξυγχρονίσουμε την πολιτική συνοχή, να την κάνουμε ένα πιο ε, απλό και αποτελεσματικό ε, χρηματοδοτικό μέσο. Χρειαζόμαστε ε, μέσα όπως το Τζέρεμι, το Jasper και το Τζέσικα μηχανισμούς ανακύκλωσης, δηλαδή όπου τα χρήματα που λαμβάνει ο δικαιούχος επιστρέφονται και ξαναδαπανώνται για άλλα προγράμματα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει πολύ πιο ολοκληρωμένος προγραμματισμός. και οι δράσεις να βασίζονται σε αυτόν. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση σε όλα αυτά τα σεμινάρια ήταν ο τρόπος είναι ότι κάποια πράγματα που λέμε είναι τελείως ακατανόητα. Άλλα λέμε στις Βρυξέλλες, άλλα λένε στις ε, πρωτεύουσε, άλλα λένε στις περιφέρειες, άλλα ακούμε στα χωριά. Στις Βρυξέλλες πρέπει να είμαστε σαφείς. Πρέπει να εξηγούμε τι λέμε. Και έτσι ο κόσμος θα στηρίξει αυτά που προσπαθούμε να πετύχουμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχω πέντε ομιλητές ε, στον κατάλογο. Θα δώσω τρία... Πρώτα θα ακούσουμε τους ε, τρει εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Λόρδος Χάσκινς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Καταρχήν, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά το, το διαθέσιμο ποσό χρημάτων. Μιλάμε για ένα προϋπολογισμό ε, που αποτελείται από το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Κάποιοι θέλουν να είναι περισσότερο, αλλά ε, το πιθανότερο είναι ότι θα παραμείνει 1%. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές. Ε, δεύτερον, Ο στόχος για τις στοχές χώρες ήταν ε, η πιο αποτελεσματική πτυχή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια και τη ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνει σημαντικό στόχος. Η κυβέρνηση της Βρετανίας πιστεύει ότι αυτό είναι σημαντικό. Τρίτον, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τομεί όπου είναι διαμφισβήτητος ο ρόλο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο ακόμα πιο σημαντικό το ευρωπαϊκό κοινό θα συμμετέχει στα προγράμματα ώστε και, εκείνη, και το κοινό να ε, συμμετέχει. Και τρίτον, χρειαζόμαστε μια πιο ολοκληρωμένη συνεκτική ε, προσέγγιση στην ενέργεια, διότι αυτό είναι κάτι που όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκτιμήσουν και θα καταλάβουν. Το θέμα τη ε, κλιματική αλλαγή ε, που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη του κοινού τα τελευταία χρόνια, είναι και αυτό ένα θέμα που θα πρέπει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο που με, που με ανισχύει εμένα πάρα πολύ, επειδή ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για την ανώτατη εκπαίδευση, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί σε σχέση τη Βόρεια Αμερική και όλο και περισσότερο σε σχέση και με την Ασία στον τομέα τη ε, ανώτατη εκπαίδευση. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ιδιαίτερα την ποιότητα τη ανώτατη εκπαίδευση που παρέχουμε στου νέου ανθρώπου. Η πέμπτη τελευταία μου παρατήρηση είναι η πιο σημαντική. Ε, μένουμε σε έναν κόσμο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για απελευθέρωση του εμπορίου, εξάλληψη των εμποδίων και τα τελευταία χρόνια. Ε, αυτή ήταν η τάση στον κόσμο. Του τελευταίου μήνε είδαμε οι τάσεις αυτές να αντιστρέφονται με καταστρεπτικές ε, συνέπειες. Και η δική μου χώρα και άλλες ε, είναι ένοχες ε, για τις προστατευτικές τους τάσεις. Έτσι θα διακυβεύσουμε όμως όχι μόνο την σύγκληση αλλά και το όλο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διακυβευτεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. από τον Nationalrat της Αυστρίας, ο κύριος Στάτλερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ με τον Πολωνό συνάδελφο ότι δεν έχει νόημα να πανικοβληθούμε λόγω της ε, λόγω της ε, κρίσης, αλλά και ε, ε, εξοραίζοντάς την πάλι δεν πετυχαίνουμε τίποτα ανησυχώ ότι οι συνέπειες της ε, κρίσης και συμφωνώ με τον ε, Ούγγρο συνάδελφο μετά το έτος 2013 δεν θα έχουν ξεπεραστεί. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει η κρίση, αλλά οι συνέπειες της κρίσης αυτής ε, θα μας απασχολούν και μετά το 2013. Θα δούμε αυξανόμενη ανεργία θα αντιμετωπίσουμε ανεργία τέτοιου μεγέθους που ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε πριν ε, κάποια χρόνια. Ήθελα απλά να τονίσω αυτό που είπαν οι συνάδελφοι από την Ιταλία και την ε, ε, Ισπανία. Θα δούμε μαζική ανεργία, νέο φαινόμενο πολύ μεγαλύτερου μεγέθους και ιδιαίτερα όσον αφορά την ανεργία των νέων μας έχουν τρομάξει αυτά που συνέβησαν στην Αθήνα την τελευταία εβδομάδα και έχουμε με την ανεργία το πρόβλημα της κοινωνικής ειρήνης. Λύση δεν μπορεί να είναι ε, να καθόμαστε και να κοιτάμε την ανεργία να αυξάνεται και να βλέπουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Έτσι όλοι οι στόχοι που είχαμε θέσει τα τελευταία χρόνια στην περιφερειακή πολιτική θα ε, εξαφανιστούν. Θα πρέπει να αντισταθούμε σε μια τέτοια εξέλιξη. Δεν ε, νομίζω ότι υπάρχει πιο σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή από την καταπολέμηση της ανεργίας. Ο στόχος της πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να είναι κοινό ευρωπαϊκό στόχο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, των κρατών μελών αλλά και τη περιφερειακή πολιτική. Η κοινωνική ειρήνη στι χώρε μα θα εξαρτάται τα επόμενα χρόνια από το αν καταφέρουμε να διασφαλίσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν την πλήρη ε, απασχόληση. Εάν δεν το πετύχουμε, ο κόσμο δεν θα ικανοποιηθεί με στόχου που αφορούν την, αφορά, την αλλαγή του κλίματο. Θα μας ε, ρωτήσουν πότε θα έχω δουλειά, όχι πότε θα αλλάξει το κλίμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάθε πρόγραμμα στο μέλλον, ιδιαίτερα στον τομέα τη ε, περιφερειακή πολιτική θα πρέπει να εξεταστεί ανάλογα με τις συνέπειες του στην ε, απασχόληση, στην ε, καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, στην καταπολέμηση της ανεργίας των γυναικών και στην ε, καταπολέμηση της ανεργίας για ανθρώπους ηλικίας άνω των 50 ετών. Αυτοί οι τρεις τομείς έχουν ιδιαίτερη συμφωνία. Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να εξεταστεί υπό το φως της ε, καταπολέμησης της ανεργίας και της ε, διασφάλισης της πλήρους απασχόλησης. Δεν είμαι αφελής ώστε να πιστεύω ότι με την ε, περιφερειακή πολιτική και μόνο θα πετύχουμε την πλήρη απασχόληση. Αυτό δεν το πιστεύει κανείς. Όμως η πολιτική αυτή των μεμονωμένων κρατών μελών, η περιφερειακή πολιτική, και συνεχώς και η πολιτική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ε, πολιτικής συνοχής θα πρέπει να στοχεύουν ακριβώς εκεί. Δεν θα υπάρχει κατανόηση στα κράτη-μέλη εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιφερειακή πολιτική της ε, διατυπώσει άλλο κεντρικό σημείο από ότι αυτό που θα πρέπει να ε, διατυπώσουν τα ε, κράτη-μέλη ως ε, κεντρικό θέμα, την καταπολέμηση της ανεργίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με το θέμα αυτό. Όλα τα άλλα προβλήματα είναι μεν σωστά, αλλά αλλά σε σχέση με, το, ε, με τη διασφάλιση ε, ε, μέσων ζωής για τους ανθρώπους μάλλον είναι δευτερεύοντα. Και τέλος ο κύριος Φερνάντης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ένα θέμα που όλου μας ενώνει εδώ είναι η πολιτική συνοχή και αποτελεί και στοιχείο του ευρωπαϊκού DNA, της ευρωπαϊκής ηθαγένειας και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. η Ευρωπαϊκή Συνοχή δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπει στο χρονοτούλαπο. Θα πρέπει να ενισχυθεί και να συνεχιστεί. Μίλησε ο κύριος Γκελέκ για την τέταρτη έκθεση συνοχής, για την έκθεση Άλενμπαχ και τα λοιπά και αύριο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας για τις καλές πρακτικές της περιφερειακής πολιτικής. Όλα αυτά για μένα δείχνουν ότι το Κοινοβούλιο θέλει να συνεχιστεί η πολιτική αυτή. Η σημερινή λοιπόν συνεδρίαση θα δώσει κάποια μηνύματα και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν να συνεχίσουν ε, την πολιτική αυτή, θέλουν να συνεχιστεί η πολιτική και αυτό διατρανώνουν και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής φαίνεται γιατί είναι πολλοί οι πολίτες και πολλά τα κράτη που θέλουν να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τα λέω αυτά. Δεν τα λέω αυτά επειδή είμαστε προεκλογική περίοδο που είμαστε και αυτό σημαντικό είναι, αλλά το πρόγραμμα αυτό της συνοχής είναι μακράς πνοής ε, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και οικοδόμησης. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς θέλω να σας υποβάλω μερικές σημειώσεις. Και να πω πρώτον, αυτή η συνάντηση ήταν πάρα πολύ θετική. Καλό θα ήταν κύριε Πρόεδρε ε, τα κοινοβούλια των κρατών μελών να οργανώνουν τέτοιες ε, συναντήσεις, τέτοιες διασκέψεις στις χώρες και στις περιφέρειες που έχουν και κοινοβούλια. Όπως είπε προηγουμένως μια συνάδελφος, με εκπροσώπους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δήμων και των κοινοτήτων. Επιτρέψτε μου να σας πω τα εξής λοιπόν. Η, αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά ε, από τη χρηματοδότηση. Καταρχήν δεν θα πρέπει να γίνει επανεθνικοποίηση. Συνεργασία χρειάζεται των διαφόρων επιπέδων πολιτικής από την ευρωπαϊκή μέχρι ε, το εθνικό επίπεδο και το περιφερειακό. Έχει δίκιο ο κύριος Πανιστερόη που λέει ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή θεώρηση. Αλλά επίσης δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έχει και ιδιαίτερες περιφέρειες με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, νησιωτικές περιοχές ας πούμε ή ε, αραιοκατοικημένες περιοχές. Και εγώ προέρχομαι από μία άκρος απομακρυσμένη περιφέρεια και τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα. Φέρνουν στην Ευρώπη νέα διάσταση και είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουν υπόψη και οι δικές τους ιδιαιτερότητες. Ένα άλλο στοιχείο ε, που ανέφερε η Τσεχική Προεδρία είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό της πολιτικής συνοχής με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές είναι απολύτως απαραίτητο να ενισχυθεί η πολιτική συνόχη από το 2013, οπωσδήποτε. Και τελειώνω, γιατί βλέπω το σφυρί να με απειλεί. έλεγα λοιπόν ότι η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να δώσει νέα όθηση και γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη συνθήκη και γι' αυτό ε, αξιοποιώ και, και εκμεταλλεύομαι την τσεχική προεδρία για να πω ότι Ε, γίνονται πολλές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε και να αφήσουμε τα πράγματα να πάρουν την πορεία τους, αλλά και η Τσεχική Προεδρία να συνεισφέρει και το Τσεχικό κράτος ε, όπως το αναλογεί και αυτό θα γίνει με την έγκριση της συνθήκης και απευθύνω έκκληση. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Λούιτσι Λούζι, τελευταίος εθνικός βουλευτής και συγκεκριμένα γερουσιαστής από την Ιταλία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η νέα πολιτική συνοχή επέτρεψε να επανακαθοριστούν οι προτεραιότητες των κρατών μελών για την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την κοινωνία της πληροφορία κτλ. Είδαμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αξιοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά έχουν ενισχυθεί και βλέπουμε και μια νέα ορολογία να χρησιμοποιείται, ένα νέο λεξιλόγιο που ήρθε να πλουτίσει το ευρωπαϊκό λεξιλόγιο χωρίς να ε, αδειάσει από ουσία η συνοχή με την αηφόρο ανάπτυξη, με την αλληλεγγύη. Αλλά ε, τώρα έχουμε νέες ε, προκλήσεις. Έχουμε μια νέα προγραμματική περίοδο, ένα νέο κύκλο και θα πρέπει να συνδεθεί η στρατηγική της Λισαβόνας με τη πολιτική συνογής. Τα κράτη-μέλη το γνωρίζουν αυτό και το καταλαβαίνουν. Δεν θα πρέπει όμως η στρατηγική της Λισαβόνας για τους στόχους τους να αντλήσει κονδύλια από τα ταμεία συνοχής σε καμία περίπτωση. Δεν θα πρέπει να λισαβονοποιήσουμε την πολιτική συνοχής. Δεν θα βοηθήσει αυτό. Εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις ε, του μέλλοντος. Ε, καλή στρατηγική της Λισαβόνας έχει εξυγχρονιστεί, έχει ανανεωθεί με νέους στόχους, αλλά παραμένουν οι στόχοι αυτοί πολύ γενικόλογοι και αόριστοι και κινδυνεύουμε να χάσουμε κοινοτικούς πόρους, να διαχυθούν τα κεφάλαια προς κατευθύνσεις πολύ αόριστες και αυτό είναι κρίμα και θα ήταν εις βάρος της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να έρχεται από τις περιφέρειες σε συνεργασία με τα κρατημέλη και τελικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να χαράσετε με τρόπο ε, που να σέβεται και αυτή τη χωρική territorial διάσταση και να ε, γράφονται όλα αυτά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος για την Ανάκαμψη της Οικονομίας. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε σε αυτή την περίοδο κρίσης να προχωρήσουμε και είναι πολύ σοβαρή η κρίση γιατί περνάμε από την ύφεση σε ένα πραγματικό κράκ, σε ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση της οικονομίας. Δεν είναι ύφεση, είναι κράκ, λοιπόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περιορισμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο σε κάποιες δαπάνες. Δεν ισχύει αυτό για τις διαρθρωτικές δαπάνες. Στα πλαίσια όμως της συναπόφασης θα μπορεί να ε, ελέγχει περισσότερο και τα δημοσιονομικά. Και τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στα σημαντικά θεμελιώδη ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί περίπου 65% στην πολιτική συνοχή μάλλον αφιερώνει το 65% ε, των κοινοτικών κονδυλίων του κοινοτικού προπολογισμού. Θα πρέπει και μετά το 2013 να ενισχύεται αυτή η πολιτική και να αποκρούσουμε κάθε απόπειρα επανεθνικοποίησης που επιχειρούν ορισμένα κράτη-μέλη. Δυσκολίε υπάρχουν, αλλά η πολιτική συνοχή έχει αποδείξει ότι κατάφερε να προσαρμοστεί στις ε, δυσκολίες. Η κρίση χρειάζεται ειδικέ απαντήσεις σήμερα και επιλογές για το μέλλον. Θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, όπως είπε ο κύριος Άνερ, Γενικός Διευθυντή ε, στην εισαγωγή του, και θα πρέπει να απλουστεύσουμε και τις διαδικασίες ε, της συνοχής στη διαχείριση των κονδυλίων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω, να σας χαιρετήσω με μια συγκεκριμένη πρόταση. Να μπορέσουμε να συζητήσουμε για την χρήση των διαρροτικών ταμείων ε, στο πλαίσιο ενός επίσημου ε, Συμβουλίου των Υπουργών να προβλεφθεί δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ε, τυπικό βήμα για εμβαθυμένη πολιτική συζήτηση που ακόμα λείπει για την πολιτική του 2013 και μετά. Σας ευχαριστώ. Τελευταίοι δύο μιλητές, σύντομες παρατηρήσεις παρακαλώ από τον Γενικό Διευθυντή και συμπεράσματα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεράρντο Γκαλεότε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το ότι μπορέσαμε να έχουμε αυτή την συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Θα πρέπει να σας πω ότι θα γυρίσω στο σπίτι μου με πολύ τροφή προσκέψη, όχι μόνο για απόψε το βράδυ, αλλά <laughs> για τις επόμενες εβδομάδες νομίζω. Επίσης να ευχαριστήσω πολύ όλα τα μέλη για την ενθάρρυνση την οποία μου έδωσαν όσον αφορά την περαιτέρω εξέλιξη της πολιτικής συνοχής. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για να αποφευθεί η παρεξήγηση για κάτι που είπα στην αρχή και να πω και δύο λόγια για την πολιτική συνοχή στο πλαίσιο της ε, τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Θα έλεγα, ε, είπα καταρχήν ότι στην αρχή ότι στο μέλλον θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε στο, πλαίσιο, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής περισσότερη ε, μέσα πιστοτικής ε, μηχανικής. Μέχρι στιγμής δουλέψαμε με, με, επιδοτήσεις, δηλαδή δίναμε επιδοτήσεις και από τη στιγμή που δίνονταν οι επιδοτήσεις τελείωσε. Στο μέλλον πιστεύουμε πως ε, τουλάχιστον σε τμήματα της πολιτικής μας υπάρχουν επενδύσεις όπου δεν είναι απαραίτητα ο καλύτερος τρόπος και ο πιο αποτελεσματικός ε, τρόπος να δώσουμε επιδοτήσεις ή χορηγίες, δηλαδή επενδύσεις που μπορεί μετά να γεννούν εισοδήματα, μπορεί να αξίζει τον κόπο να μην δίνουμε επιδοτήσεις αλλά να τις χρηματοδοτούμε μέσω πιστοτικών μηχανισμών. Και αυτό είναι το τμήμα του πιστοτικής ε, μηχανικής που σας είπα. Η μεγάλο πλονέκτημα είναι τα δημόσια χρήματα δίνονται για στήριξη αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές και να είναι πιο αποτελεσματικά. Επίσης θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν μπορούν όλα να χρηματοδοτηθούν όλα με αυτόν τον τρόπο. Πιστώσεις για παρά... Ε, ε, επίσης, κατά την άποψή μας, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Η πρόσβαση στην πίστοση έχει γίνει εξαιρετικά ε, δύσκολη λόγω της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης και το βλέπουμε και στην πολιτική μας διότι αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα η ζήτηση για τα προγράμματα Jeremy και Jessica που υπάρχουν ήδη πίστοση λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την οικονομική επιβίωση των μικρομεσαίων μας επιχειρήσεων. Κάποιες φορές όμως ακόμα και των μεγάλων επιχειρήσεων. Η συμβολή της πολιτικής συνοχής στην επίλυση της κρίσης μπορεί, και αυτό το λέω με κάθε ειλικρίνεια, μπορεί να είναι μόνο μέτρια για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σε σύγκριση με τα μέτρα κατά της κρίσης που θέτουν σε εφαρμογή τα κράτη-μέλη μας είναι μια στάλα σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με αυτά τα μέτρα. Μιλάμε για 30 δις ετησίως, νομίζω 24 δις για το 2009, 30 δις ετησίως σε σύγκριση με τα αντικυκλικά προγράμματα που έχουν αναπτύξει ορισμένα από τα κράτη-μέλη μας. Αυτά είναι πολύ λίγα. Αλλά επίσης η πολιτική συνοχή έχει στόχο και νομίζω θα πρέπει να παραμείνει έτσι μια διαφορετική πολιτική. Δηλαδή αυτό σημαίνει μια πολιτική που διατηρεί μια πιο μακροπρόθεσμη οπτική για το πού θα πρέπει να, θα πρέπει να είναι η στόχη μας στην ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί ένα στοιχείο συνέχειας και σταθερότητας. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που βλέπουμε κάποιες φορές σε καταστάσεις κρίσης είναι ότι οι επενδύσεις στους στρατηγικούς τομείς για το μέλλον όπως η παιδεία, η ανώτατη εκπαίδευση, η έρευνα και ανάπτυξη, η καινοτομία είναι πολύ συχνά ε, μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο λόγω άλλων επιγόντων αναγκών. Η πολιτική συνοχής ανέκαθεν στους στόχους της συμπεριλαμβάνει και το στόχο της απασχόλησης και νομίζω πως θα είναι ένας πολύ πολύ σημαντικός ε, στόχος για τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια και πέρα από το 2013 και όχι μόνο με σχέση με αυτή την κρίση αλλά ενισχύεται σε αυτή την κρίση. Πολύ η κατάσταση. Αν δούμε σε περιφερειακή ανάλυση έχουμε περιφέρειες στην Ευρώπη όπου θα έχουμε πραγματικά προβλήματα ανεργίας, ανεργίας ενώ ταυτόχρονα στο μέλλον μπορεί να έχουμε απερίμωση σε κάποιες άλλες περιφέρειες. Δηλαδή, περιφέρειες όπου έχουν, τις έχουν καταλήψει οι νέοι και έχουμε μια πολύ γρήγορα γυράσκουσα κοινωνία. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να λυθούν μόνο ε, μέσω πολύ σοφά συνδυασμένων πολιτικών. Χρειαζόμαστε πολιτικές που θα εξετάζουν τη συγκεκριμένη περιφερική κατάσταση και που θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν απαντήσεις από, για τη συγκεκριμένη περίπτωση κάθε φορά, που θα αντιστοιχούν, θα αντιστοιχεί δηλαδή στη συγκεκριμένη περιφερική περίσταση. Και αυτό είναι ένα σημείο ένας λόγος μάλλον για τον οποίο το πρότυπο της πολιτικής συνοχής που έχουμε όπου αναπτύσσονται προγράμματα σε περιφερειακό και κάποιες φορές σε εθνικό επίπεδο και έπειτα ανεβαίνουν ε, παραμένει πολύ σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σταματήσω γιατί υπάρχουν τόσα πολλά που θα μπορούσα να πω. Ελπίζω μόνο ε, ότι θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εξαιρετικά πλούσια συζήτηση και ότι θα μπορέσουμε και μάλλον να κλείσω ευχαριστώντας την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διοργάνωσε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ε, ε, βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενικέ, σε μένα έπεσε ο κλήρος να ολοκληρώσω αυτή την πρώτη συνεδρίαση των Επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι μια πρωτοβουλία που ε, χαρακτηρίζεται από την ενισχυμένη εξουσία που δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας στα Εθνικά Κοινοβούλια στη νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελπίζω να συμφωνήσουν όλα και τα ε, εθνικά κοινοβούλια είναι τέτοιου είδους συνεδριάσεις να παγιωθούν. Και διαλέξαμε ως θέμα της πρώτης αυτής συνάντησης στο μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2013. Γιατί ούτε δύο χρόνια δεν έχουν περάσει. Μόλις δύο χρόνια πέρασαν από τη θέση ισχύ των ισχυουσών δημοσιονομικών πρόπτικων και ήδη από τώρα εργαζόμαστε για να προετοιμάσουμε το μέλλον. Και όπως επανειλημμένα ακούστηκε εδώ κατά τη διάρκεια του απογεύματος σήμερα, η οικονομική κρίση που μας πλήττει κατέστησε σαφές ότι το πιο ισχυρό κοινοτικό μέσο, ίσως και το μόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε οικονομικά είναι η πολιτική συνοχής. Όσο μετριοπαθής και να είναι η χρηματοδότησή της και η συνεισφορά. Τις προτάσεις ε, και τα συμπεράσματά μας που θα συντάξει η γραμματεία μας θα τις διάσουμε στη συνέχεια και κανονικά εγώ θα επιθυμούσα ε, να σας τις ε, παρουσιάσω σε πολλές, κάποιες πενελιές, αλλά μου λένε ότι είστε υποχρεωμένοι να φύγετε πολύ γιατί έχετε πτήσεις να πάρετε. Οπότε, απλώς θέλω να σας πω ότι θα σας στείλουμε τα συμπεράσματά μας και τις προτάσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας μόνο ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η πολιτική συνοχής είναι η πλέον ορατή και η πλέον επιτυχής από όλες τις κοινοτικές πολιτικές. Και αυτό ισχύει. Όχι μόνο για τις χώρες και τις περιφέρειες της συνοχής, αλλά και για τους καθαρούς συνεισφορείς τους λεγόμενους. Διότι σε τελική ανάλυση επωφελούνται όλοι από την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πολιτική συνοχής που μέχρι τώρα αποτελούσε σημαντικότατο πυλώνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αυτό τον καιρό λοιπόν δείχνει ακόμα περισσότερο η πολιτική συνοχή και πλήρως πόσο ισχύει στο ακέραιο και η συνεισφορά της από το έτος 2013 και μετά βεβαίως με τις απαραίτητες προσαρμογές ε, στη πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ε, ζωτική σημασίας. Επίσης ακούστηκε και αυτό και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη που όλοι προσδοκούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω ότι θα σας στείλουμε τις προτάσεις και τα συμπεράσματα και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε στην επόμενη συνάντηση που όλοι δεσμευτήκαμε να διοργανώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.